Good morning. Please use for your headphone. I am speaking Spanish. Bueno, pues eh, empezamos. Repito, buenos días a, a todos y a todas. Λοιπόν, σας καλωσορίζω όλους. Θα ξεκινήσουμε με την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν. Ο κύριος Χάουτ είναι ο εισηγητής μας. Έχουν κατατεθεί άνω των 400 τροπολογιών και υπάρχουν 26 συμβιβαστικές προτάσεις. Δίνω το λόγο στον κύριο Χάουιτ. Uh, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε θα συγκεντρώσω την προσοχή μου στις συμβιβαστικές ε, προτάσεις τις οποίες έχουμε διαπραγματευτεί σήμερα. Ξέρετε ότι υπάρχουν έντονες απόψεις στο Κοινοβούλιο και στις πολιτικές ομάδες γύρω από το θέμα αυτό. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους οι οποίοι πήραν μέρος στην προσπάθεια που έγινε για τις συμβιβαστικές. Να πω ότι η Επιτροπή μας Ε, στην Επιτροπή μας ότι δεν είναι κατεπήγον το θέμα, ε, δεν είναι αν θέλετε μια έκθεση γενικά για το Ιράν, να μην υπάρχει παρεξήγηση εδώ. Δεν είναι μια συναλλική έκθεση για το τι συμβαίνει στο Ιράν. Ε, ούτε είναι κάτι το οποίο ασχολείται ειδικά με το θέμα των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ιράν έχει ένα συγκεκριμένο θέμα και αυτό το λάβαμε υπόψη μας όταν διατυπώσαμε τις συμβιβαστικές. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να έχουμε μία έκθεση η οποία να είναι επικοδομητική και να μας βοηθήσει στο στόχο μας να επανέλθει το Ιράν στην διεθνή ε, τάξη. Να είναι τμήμα της διεθνούς ενόμου τάξεως το Ιράν. Αυτό για μας είναι καθοριστικό, είναι σημαντικό. Φυσικά η συμφωνία αυτή θα πρέπει να είναι δίκαιη και η έκθεσή μας θα πρέπει να είναι δίκαιη, να σέβεται τις διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι τομείς όπου οι συνάδελφοι, κάποιοι εκλεκτοί συνάδελφοι θεώρησαν ότι δεν ήταν απόλυτα ισορροπημένη η έκθεση και γι' αυτό ακριβώς προσπάθησαν να καλύψω τις ανησυχίες Λοιπόν, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας να ασχοληθώ με όλα αυτά επιμέρους αν θέλετε. Στο 1 και στο 3 κάνουμε ειδική αναφορά στον ρόλο της είπα της εκπροσώπου. Γίνεται συγκεκριμένη αναφορά και για την ανάγκη στήριξης της προσπάθειας την οποία έχει ξεκινήσει η, η Υπηρεσία Εξωτερικών Θέσεων. Ζητήσαμε επίσης τη δημιουργία και μιας αντιπροσωπείας με το Ιράν και τέθηκε εδώ το θέμα των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σαφές ότι στην Τεχεράνη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σωστή αντίληψη για τον ρόλο τον οποίο παίζουν τα θεσμικά όργανα και γι' αυτό όταν πήγα στην Τεχεράνη Προσπάθησα να πιέσω τους συναδέλφους εκεί και να τους πω ότι είναι βασικό να δουλέψει η αντιπροσωπεία. Δεν είναι θέμα δημοσιονομικό ή μια απόφαση εδώ σε εμά, αλλά νομίζω ότι και αυτοί πρέπει να πάρουν την κατάλληλη απόφαση για την λειτουργία της διακοινοβουλευτικής. Για τη συμβιβαστική 7 αφορά την διαφάνεια, την ελεύθερη αγορά και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα μας ενδιαφέρει ανεξαρτήτως πολιτικών καταβολών του καθενός. Εμείς θέλουμε μια τέτοια συμφωνία να μπορέσει να δουλέψει και γι' αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το Ιράν έχει αναλάβει στα πλαίσια του προγράμματος δράσης ε, ορισμένες υποχρεώσεις Πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν την προσπάθεια αυτή και να δούμε ακριβώς τι μέτρα θα ληφθούν στον τομέα της ολοκλήρωσης της ελεύθερης αγοράς και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Υπάρχει επίσης και ένα άλλο θέμα αρκετά δύσκολο για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό είναι κάτι το οποίο τίθεται σε συζήτηση κάθε φορά που πηγαίνει κάποιος εκπρόσωπος χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ε, ε, Ιράν, κάθε φορά που πηγαίνει κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τίθεται το θέμα των κυρώσεων Ξέρετε ότι υπάρχει ένας κάποιος αντιαμερικανισμός και στην Τεχεράνη και σε πολλές άλλες χώρες και γι' αυτό εμείς προσπαθήσαμε με έναν τρόπο ο οποίος ελπίζω θα μπορέσει να βοηθήσει να βρεθεί ε, μια λύση, ιδιαίτερα στη συμβιβαστική δέκα. Νομίζω ότι είναι, υπάρχουν κάποιες εμπορικές συμφωνίες οι οποίες ε, ε, εφόσον ολοκληρωθούν είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν τη βελτίωση του κλίματος. Τώρα για το περιβάλλον συμμερίζομαι τις ε, προτάσεις που έχουν γίνει. Θέλουμε να υπάρξει συνεργασία στον τομέα της ενέργειας And it is a concern that I have, and so I've been very happy to adopt that element of Mr. Bruckner's amendment. And I did have a very good meeting in Tehran with civil society. Λοιπόν, επίση θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε επαφές και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, να αναπτύξουμε λοιπόν τις σχέσεις αυτές στο Ιράν, κάτι το οποίο θα το δείτε στις τροπολογίες 11 και 12, τις συμβιβαστικές. Για το 2013 χρειάζεται επίσης ε, να υπάρξει διάλογος για τα θέματα της μετανάστευσης, όπως υπάρχει ένας αντίστοιχος τέτοιος διάλογος ε, με άλλες χώρες. Απαιτείται να υπάρξει ένας τέτοιος διάλογος. Στο 2014 είχα επισκεφθεί συγκεκριμένα το Πανεπιστήμιο στην Τεχεράνη τεχνική βοήθεια, επιστημονική συνεργασία στον τομέα της έρευνας και ανταλλαγές σε φοιτητικό επίπεδο, σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Είναι μια καλή ευκαιρία για όλους και για μας εδώ στην Ευρώπη. Στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βέβαια ε, το θέμα μας δεν είναι κατεπήγον, αλλά πρέπει να είμαστε σωστοί και δίκαιοι ξεκαθαρίζουμε εδώ το θέμα ότι πρέπει να μειωθεί το φαινόμενο δυστυχώς αυτό της ε, θανατικής ποινής και πρέπει να σταματήσουν ε, όλες ε, οι εκτελέσεις issues, freedom expression, of course, that end up Πρέπει λοιπόν να βρεθεί κάποιος κοινός στόχος εδώ θα δείτε στις τροπολογίες που έχουν κατατεθούν για την θανατική ποινή ότι ξεκαθαρίζουμε ότι είμαστε υπέρ της κατάργησης και ζητούμε να εφαρμοστεί αμέσως ένα μορατόριο άμεσα. Σχετικά τώρα με τις σχέσεις Ιράν-Σαουδικής Αραβίας, συμβιβαστική 16, ζητάμε από τις δύο αυτές χώρες ε, να μην προβαίνουν σε επιθετικές ενέργειες ε, και να μην υποστηρίζουν εχθρικές ένοπλες ομάδες στην περιοχή. Βλέπετε ότι η διατύπωση αυτή είναι πάρα πολύ προσεκτική αλλά και δίκαιη σε σχέση με τις δύο πλευρές. Στοχεύουμε λοιπόν και τη Σαουδική Αραβία αλλά και το Ιράν. Ονοματίζουμε τις χώρες αυτές αν θέλετε. Ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο, είμαι συνοπτικός. Σχετικά η συμβιβαστική πρόταση τώρα για τις εκλογές και την εξέλιξη των δημοκρατικών θεσμών στο Ιράν. Εδώ είναι ένας τομέας στον οποίο οι, οι συνάδελφοι ήθελαν να υπάρξουν αρκετές αλλαγές. Ε, προχωρήσαμε στις αλλαγές αυτές Είχαμε μια μακρά συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό ήδη στο παρελθόν και ελπίζω στα πλαίσια της συζήτησης αυτής να υπάρξει υποστήριξη. Για το 22 εμείς υποστηρίζουμε τους ειδικούς μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράν Νομίζω ότι η ρητορική την οποία χρησιμοποιούμε είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει δεκτό και σε τομείς όπως ο σεβασμός των θρησκευτικών ελευθεριών, ο σεβασμός των μειονοτήτων, Ελπίζω επίσης και στα θέματα των δικαιωμάτων των γυναικών, στο θέμα του γενετήσιου προσανατολισμού, Πρόκειται για τη συμβιβαστική 25, αν δεν κάνω λάθος. Ελπίζω να είναι ισορροπημένη. Νομίζω ότι άκουσα τους συναδέλφους αυτό το οποίο ζήτησαν. Ελπίζω να μείνουμε στα όρια τα οποία θέτει η έκθεση αυτή φιλοσοφία της έκθεσης αυτής δεν είναι να βάλουμε μέσα ό,τι θέλει ο καθένας ή ό,τι πιστεύει ότι είναι σωστό ο καθένας. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βάλουμε κάποιες κοινέ θέσεις οι οποίες να είναι θέσεις που θα επηρεάσουν την εξέλιξη των πραγμάτων στην Τεχεράνη. Αυτή είναι η σημασία της συγκεκριμένη έκθεσης και θα πρέπει σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξουμε τις διαδικασίες που έχουμε επιλέξει. Ευχαριστώ κύριε Χάουιτ για την εργασία σας. Ποιος? Ο κύριος Αντάκτουσον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συμμετείχα Εξ αρχής, ε, έχοντας μεγάλες ανησυχίες σε, αυτό το, αυτή την πρόταση ψηφίσματος, 2.500 ε, λέξεις είναι στο πρωτότυπο, αλλά τρεις φορές μόνο αναφέρονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, είμαστε επικριτικοί για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τα στερεότυπα. Ε, δεν καταδικάζουμε ούτε μία φορά τη, μία από τις πλέον κτηνώδεις δικτατορίες. Βρισκόμαστε σε πλήρη αντίφαση με τις λέει ανησυχητικές εκθέσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Από την Amnesty International η έκθεση αναφέρει πως ε, η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν επιδεινώνεται σταδιακά και δεν ε, φαίνεται στον ορίζοντα καμία δυνατότητα βελτίωσης. Η δικτατορία αυτή διώκει τους πολίτες του Ιράν και παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πέραν αυτού, αυτό το καθεστώς όπως ξέρουμε υποστηρίζει το Χεσμολά και τη Χαμάς ε, και άλλες ε, παρόμοιες ε, τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι κράτος τρόμου και είναι υπεύθυνη για κατεξοσιοδότηση πολέμου στην Συρία, στο, στην Ιεμένη. Ευθύνεται το Ιράν για την ανίποτε δυστυχία χιλιάδων αθώνα μάχων. Τίποτα από όλα αυτά, συνάδελφοι, δεν αναφέρεται στην έκθεσή μας. Η υπογραφή της πυρηνικής συμφωνίας τι σημαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι είναι αξιόπιστος εταίρος του Ιράν. Προσοχή. Πρόσφατα διάβασα στο Economist ένα άρθρο όπου εκφράζονταν σοβαρές ανησυχίες για την Ισλαμική Δημοκρατία. Παραθέτω. Αυτοί που ήλπιζαν ότι με την υπογραφή της πυρηνικής συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις μεγάλες δυνάμεις θα ενισχυόταν ε, το κίνημα των μεταρρυθμιστών της χώρας ε, το βάρος ε, των θρησκόληπτων συντηρητικών θα έπρεπε να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους. Τέλος παράθεσης, υπάρχουν φυσικά θετικές αλλαγές που έχουν γίνει στο σχέδιο, όμως δεν επαρκούν. Έχω υποβάλει και συνυπογράψει με συναδέλφους ε, τροπολογίες που ξεκάθαρα τονίζουν πόσο σημαντικό είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι στο πυρήνα των σχέσεών μας με το Ιράν. Κλείνοντας, θέλω να πω πως ο Ιρανικός λαός χρειάζεται και αξίζει την υποστήριξή μας στον αγώνα του για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριος Μπρόκ. Ευχαριστούμε. Είμαστε στη, στο στάδιο της εξέτασης των προτάσεων. Δεν είναι η τελευταία φορά που συζητούμε το θέμα. Θα προχωρήσουμε. Μετά τις συζητήσεις των σκιωδών για το ζήτημα, οφείλω να πω πως οι προτάσεις του κ. Χάρτη για τις συμβαστικές έχουν τροποποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Οι θεμητές ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν πλέον ληφθεί υπόψη. Θανατική ποινή και ε, γενικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα. πάνονται υπόψη. και σκιώδης για το ΕΛΚ και έχω και εγώ κάθε συμφέρον να ακολουθήσουμε τη σωστή κατεύθυνση. Ο κύριος Τάνο. Um, been... Δεν συνδιαφωνώ με τίποτα από αυτά που ακούσαμε για το καταστροφικό ρεκόρ του Ιράν, τη Ισλαμική Δημοκρατία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και είμαι γνωστό επικριτή, φοδρό επικριτή εδώ και 17 χρόνια των Μουλάδων. Από τότε που άρχισα την καριέρα μου εδώ στο Κοινοβούλιο. Σημειώθηκαν κάποιες ίσονο σημασίας εξοραϊστικές ε, βελτιώσεις ε, για να καθησυχάσουν ε, τους διεθνείς επικριτές και για να ευθυγραμμιστεί το Ιράν με τις διεθνείς υποχρεώσεις του για διάφορες ε, συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει υπογράψει, παρότι επιφυλάσσεται κάθε φορά και λέει δεν είναι, εφαρμο... εφαρμοστές οι διατάξεις αν αντιτίθεται στη Σαρία ή ε, στο... στους νόμους της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Υπήρξαν κάποιες αλλαγές. Την τελευταία δεκαετία είχαμε το μορατόριο, παραδείγματο χάρη, για το λιθοβολισμό ε, ως το θάνατο των γυναικών παρότι από ό,τι βλέπω είναι, δεν είναι σαφή τα πράγματα για το μορατόριο γιατί συναντήθηκα με την ομάδα της Διεθνής Αμνηστίας ε, για το Ιράν και μου ανέφεραν φρικτά, φρικτές περιπτώσεις. Δεν χορηγούν ιατρική περίθαλψη για πολιτικούς ε, κρατουμένους, ε, για ναρκωτικά εκτελούν ανήλικους και συνεχίζουμε τη θανατική ποινή για τα σεξουαλικού χαρακτήρα πτέσματα, μοιχεία παραδείγματος, χαρέτσι τα ονομάζουμε, ε, καταλαβαίνω αυτά που λέει ο Χαντή και ε, με τους εχθρούς σου πρέπει να ε, βρίσκεσαι σε ειρήνη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ε, και ελπίζω μετά το Brexit θα ακολουθήσουμε το δρόμο της Ένωσης και του ΟΗΕ. Τα τελευταία 14 ε, χρόνια ο Νίκ ε, με ένας φίλος μου, έγινε ε, αστάλη στο Ιράκ ως πρέσβης και ελπίζω να ενώσουμε τις φωνές μας με αυτές των μεταρρυθμιστών στο Ιράν και να μην πέσουμε στα χέρια των σκληροπυρηνικών. Ε, υπάρχει και υπαξιακή αναζήτηση, αν θέλετε, σε με τέτοιες εκθέσεις ε, για το Ιράν. Ε, δύο ώρες ήμουν με τον Ρίτσαρ και την ομάδα του χτες. Διαπραγματευτήκαμε, αλλάξαμε κάποια πράγματα. Δεν ήταν αρκετά επικριτικό το πνεύμα σε ορισμένα σημεία και δώσαμε μια όθεση προς ένα πιο επικριτικό στυλ. Πάντως, εφ' εξής, την ελπίδα μας για την αλλαγή, για την καλύτερη κατανόηση, για το διάλογο, ενισχυμένο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Ιράν για την εφαρμογή της πυρηνικής συμφωνίας. Αυτός αυτή, αυτή πρέπει να είναι η επεξίδα μας για το μέλλον και ε, να κατακρίνουμε την υποστήριξη του Χεσπολά και της Χαμάς και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων. Θα πρέπει να τους δώσουμε αυτή την ευκαιρία μας αποδείξουν το αντίθετο γιατί ελκυστική εναλλακτική δεν διαθέτουμε. Τι θα γίνει, υπήρχαν όλες αυτές ε, ε, φυλακόμενες για τα πυρηνικά και ξαναλέω είμαι επικριτής ε, του Ιράν, αλλά τι να γίνει για να... Ε, ο μόνος τρόπος για να εμποδίσουμε το Ιράν το να γίνει πυρηνική δύναμη είναι να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία και από όλους τους διάβλους αρχίσουμε πίεση ε, να, ενδεχομένως να επιστρέψουν και οι κυράσεις αν δεν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις στο να προσπαθήσουμε να έχουμε πιο εντατικό διάλογο, ε, σχέσεις με τη Δύση, περισσότερες επενδύσεις ε, και εγώ εξακολουθώ να τρέφω την ελπίδα ότι για αυτή τη μεγάλη χώρα οι πολίτες θα θέλουν κάτι καλύτερο από αυτό που ζουν σήμερα. Μπροκ, ευχαριστώ. Κύριε Σακοράφα και μετά ε, η κυρία και μετά θα ε, συνεχίσουμε επί τη βάση των συμβαστικών ε, που οποίες έχουμε καταλήξει σε αυτό το στάδιο. Ευχαριστώ και την Αυστραλ... το Αυστραλιανό κλιμάκι που κατέφτασε. Συμφωνούμε με τη διαδικασία πολύ ωραία. Κύριε Σακοράφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Χάουιτ, όλοι αναγνωρίζουμε ότι το Ιράν αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική χώρα για την ευρύτερη Μέση Ανατολή, από οικονομική όσο και από γεωπολιτική άποψη. Επίσης ότι μετά από μακριά και δύσκολη περίοδο για τις σχέσεις του Ιράν με, τους, ε, με, τους, με, τον, με τον λαό της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναπτύσσεται ένας φιλόδοξος πολυεπίπεδος διατομιακός διάλογος σε κλίμα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στη βάση της αξιολόγησης των κοινών συμφερόντων και των διαφορών κατά τρόπο που να ωφελεί και τους λαούς του Ιράν αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τον κύριο Χάουιτ για τη δουλειά που έχει κάνει για να μας παρουσιάσει μια σχετικά ισορροπημένη έκθεση και για τις συμβαστικές τροπολογίες. Εκτιμώ ότι οι προτινόμενες συμβαστικές τροπολογίες καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες για την ανάπτυξη και την διατήρηση ενός ειλικρινούς και επικοδομητικού διαλόγου, τόσο στα διαφορετικά επίπεδα που προσδοκούμε να εκφραστεί, όσο και στους τομείς για τους οποίους θέλουμε να εφαρμοστεί. Θα ήθελα ωστόσο να επισημάνω πως υπάρχουν διάφορα ζητήματα που θα επιθυμούσαμε να συμπεριληφθούν με πιο σαφή τρόπο στις συμβαστικές τροπολογίες, τα οποία για λόγους περισσότερο πολιτικών σχετισμών και όχι πολιτικής ουσίας ε, έχουν αποκλειστεί. Αρχικά θα θέλαμε μια πιο περιεκτική αναφορά σε πάγιες ανησυχίες που έχουμε εκφράσει σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, όπως παραδείγματο χάρη η ανάγκη λήψης μέτρων που να διασφαλίζουν διαδικαστικές εγγυήσεις και νομικά πρότυπα δίκης δίκης. Επίση, γνωρίζετε τη σημασία που έχει προσδώσει στο παρελθόν το Κοινοβούλιο μα στο σεβασμό του ρόλου και τη εντολή του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών καλώντα την Ιρανική κυβέρνηση να διευκολύνει το έργο του χορηγώντα του ανεπιφύλακτη θεώρηση εισόδου στη χώρα. Η πολιτική μου ομάδα θα επιμείνει σε τέτοιε τροπολογίε και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο είτε κατά τη διάρκεια τη ψηφορία στην Επιτροπή είτε στην Ολομέλειά του θα διασφαλίσει ότι θα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπούχνερ είναι ο δικός μας και ο που κολλείεται σήμερα. Μου είπε πάντως να σας μεταφέρω ότι υποστηρίζουμε την έκθεση, τη βρίσκουμε σωστή και παρακαλεί οι τροπολογίε παριθμών 362 και 483 να ψηφιστούν ξεχωριστά. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο Μπροκ. Εάν εξετάσετε ήρεμα, θα έλεγα, Πόσε τροπολογίες έχουν γίνει αποδεκτέ από πολιτικέ ομάδε για να εξασφαλιστεί μια ισορροπία, θα πρέπει να σκεφτούμε ίσω εάν θα πρέπει όντως να επιμείνουν στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες τροπολογίες δηλαδή, οι πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι είναι και ζήτημα πολύ σημαντικό για τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι και αυτή η προσπάθεια ε, να επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν για να πάυσει να προωθεί την κατασκευή πυρηνικών ε, βομβών και αυτό είναι ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν τέλει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Σύντομη παρατήρηση από εσά κύριε Σιγητά. Έχουν προσέλθει ήδη οι διακεκριμένοι προσκεκλημένοι μας, γι' αυτό θα απαντήσω πολύ γρήγορα για τον κύριο Άκουρατσον Είναι πολύ ειλικρινή η τοποθέτησή σας. Εάν δεν συμφωνείτε, εγώ υποστηρίζω πάντως την, ε, συμβαστική, τις συμβαστικές προτάσεις. Έχω να πω το εξή. Έχω ζήσει όλα τα κατεπήγοντα στο Κοινοβούλιο και με τη Διεθνή Αμνηστία τα λόγια που έχω περιλάβει στις διατυπώσεις μου είναι πάρα πολύ προσεκτικά επιλεγμένα και έχω έρθει κατ' επανάληψη σε επαφή με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο στόχος της εκθέσεως μου είναι να βελτιωθεί η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Και η προσπάθειά μου είναι να ακούσουν αυτό που λέμε. Μπορούμε να επιλέξουμε την άλλη οδό, να ε, κάνουμε, ε. να γράψουμε κάτι που μας ικανοποιεί εμάς και δεν πρόκειται να το προσέξουν καθόλου εκεί. Εγώ θέλω να διαβάσουν και να ξαναδιαβάσουν το κείμενό μας. Κανείς εδώ στο Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα διαπιστευτήριά μου σε ό,τι αφορά την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος Μπρόκ, σας ευχαριστώ πολύ. Ασφαλώς θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που να όλους. Κάπως έτσι μου λέει η διέστησή μου. Θα ήθελα τώρα να απευθύνω χαιρετισμό στην κυρία Μπίσοπ, Υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας και τον συναδελφό μας κύριο Σιόμπο, Υπουργό Εμπορίου, Τουρισμού και Επενδύσεων. Σας ευχαριστώ πολύ που προσήλθατε εδώ. Ακούτε τη μετάφραση κυρία Υπουργέ. Ναι. Ωραία. Ε, ευχαριστώ λοιπόν που ε, κάνα τον κόπο και ήλθατε να μας δείτε, βρίσκω σωστό να προχωρήσει η συνεργασία. Η εξωτερική πολιτική πλέον είναι υπόθεση γυναικών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά βλέπω και στην Αυστραλία. Αυτό είναι καλό, γιατί προσφέρουν και μια ιδιαίτερη ευαισθησία στην εξωτερική πολιτική. Οι σχέσεις μας είναι πάρα πολύ σημαντικές. Υπάρχει και η συμφωνία πλαίσιο του Απριλίου 2015, την οποία υπογράψατε εσείς κύριε Υπουργέ μαζί με την δική μας κυρία Μογκερίνη και είναι πολύ σημαντικό που υπογράφει η συμφωνία αυτή και εμείς ως Επιτροπή Εξωτερικών είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε με κάθε δυνατή προσπάθεια σε μια γρήγορη επικύρωση της συμφωνίας. Αρχίζει και η διαδικασία για την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. για να προωθηθούν οι διμερείς εμπορικές σχέσεις. Η διεθνής συνεργασία που υπάρχει ήδη με την Αυστραλία σε θέματα ασφάλειας, αντιτρομοκρατίας, ασύλου, μετανάστευσης και σε άλλους τομείς, νομίζω είναι μια θετική εξέλιξη. Μας ενδιαφέρει επίσης βεβαίως οι απειλές του ISIS και στην Νοτιοανατολική Ασία του Νταέσου. Ο χώρος της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι βέβαια τεράστιος γεωγραφικά, ωστόσο οι δεσμοί και της Αυστραλίας με τις χώρες της περιοχής αυτής είναι πολύ στενές. Υπάρχει λοιπόν απειλή και για την Αυστραλία της τρομοκρατίας που ασκεί ο Άισις και άλλοι και που απειλούν και τη δική μας σταθερότητα. Γι' αυτό και ενδιαφερόμαστε και για τα θέματα τα οποία ανεφύησαν τις τελευταίες εβδομάδες των σχέσεων των, νότιο, των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας και με την Κίνα και παρακολουθούμε προσεκτικά σε μια προσπάθεια να συμβάλλουμε σε ειρηνικές εξελίξεις. Ασφάλεια και σταθερότητα εκεί, γειτονικές σχέσεις, όλα αυτά είναι σημαντικά και από μόνα τους. Τίθεται και το θέμα της πολιτικής στο προσφυγικό. Θα θέλαμε να ακούσουμε κάτι και για τη δική σας πολιτική επί του προσφυγικού, διότι υπάρχουν και αντιμαχόμενες θέσεις στο θέμα αυτό. Αυστραλία και Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνουν νέες πρωτοβουλίες και στον τομέα αυτό. Ήδη η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Μογκερίνη, συμμετέχει σε πλατφόρμα για ευρωαυστραλιανές πτυχές της συνεργασίας. Αν θέλετε να θίξετε και το θέμα του Brexit από τη δική σας σκοπιά, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η άποψή σας. Κύριε Μπίσοπ, έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Brock, and I'm... Ευχαριστώ κύριε Μπρόκ, είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας υποδέχεται μαζί με τον συνάδελφο Στίβ Τσόμπο. Είναι μεγάλη τιμή το να μπορώ να πάρω το λόγο εδώ, γιατί ζούμε σε έναν ιδιαίτερος διασυνδεδεμένο κόσμο και οι σχέσεις ανάμεσα στα κοινοβούλια, τις κυβερνήσεις και τους πολίτες ενισχύονται από τέτοιου είδους συναντήσεις. Η γνώμη σας είναι σημαντική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τους διεθνείς εταίρους της Ένωσης όπως η Αυστραλία. Μοιραζόμαστε μαζί σας μια κοινή ιστορία, ιδέες, πεπιθήσεις, συμφέροντα επίσης και κυρίως αξίες κοινές. Πιστεύουμε στην ελευθερία, πιστεύουμε στην δημοκρατία, στο, στους κανόνες του δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ανοιχτή οικονομία, στην ανεμπόδιστη ροή κεφαλαίων και αγαθών, όλα τα πράγματα τα οποία ευνοούν την ευημερία των πολιτών μας. Και αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να προωθήσουμε και στα πλαίσια της ομάδας των 20, είμαστε μέλος της ομάδας των 20, έχουμε βιώσει 20 συνεχή έτη οικονομικής ανάπτυξης στην Αυστραλία, ακριβώς χάρη και στην απελευθέρωση του εμπορίου. Πιστεύουμε ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο όμως κόσμο τα προβλήματα αντιμετωπίζονται μέσω των σχέσεων και αυτή είναι των διεθνών σχέσεων και αυτή είναι η πορεία την οποία ακολουθούμε και γι' αυτό ακριβώς βρίσκουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικούς εταίρους στον τομέα της κοινωνίας των πολιτών, ε, της επιχειρηματικότητας κτλ. Και επίσης ε, είμαστε φυσικοί εταίροι και για την αντιμετώπιση νέων απειλών ε, στον τομέα της ασφάλειας όπως η τρομοκρατία. Η Αυστραλία έχει αποδείξει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μπορεί να δώσει κάποιες απαντήσεις. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη και εδώ στις Βρυξέλλες και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι θέματα τα οποία μας έχουν σοκάρει βαθιά λόγω της δράσης του isis νταές, όπως θέλετε πείτε του. Ε, συμμετέχουμε λοιπόν, συνεργαζόμεθα μάλλον με ομάδες ε, ε, στην Ευρώπη, με υπηρεσίες της Ευρώπης όπως τη Europol και νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά βέβαια το ίσις αν δεν υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και αν δεν σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία. Πρέπει επίσης να βελτιωθεί η ασφάλεια σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ. Ε, εμείς συνεργαζόμαστε με όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου και στα πλαίσια της καταπολέμησης του ίσης και συνεισφέρουμε στρατιωτικά και στις στρατιωτικές αποστολές της διεθνούς κοινότητας σε χώρες όπως το Ιράκ. Βοηθούμε στην, στον σεβασμό, στην τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην δημιουργία ενός κράτους δικαίου και πιο ανθεκτικών κοινωνιών. Ε, συνεργαζόμαστε επίσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Σαν παράδειγμα έχουμε τηρήσει τις κυρώσεις τις οποίες πρώτη επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα μετά από την κατάρριψη του Μαλαισιανού επιβατηγού αεροσκάφους ήταν πολύ Αυστραλοί ανάμεσα στους 300 ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με την κατάρριψη αυτή. Ο κόσμος λοιπόν γνωρίζεται ότι προσβλέπει στην Ευρώπη ε, σαν σημαντικό παράγοντα της διεθνούς τάξεως και του διεθνούς δικαίου και τον ίδιο ρόλο προσπαθούμε και εμείς ε, να αναλάβουμε στην δική μας γεωγραφική περιοχή. Θέλουμε οι κανόνες οι διεθνείς ε, να γίνονται σεβαστοί από όλες τις χώρες. Αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση σαν παράδειγμα της νότιας συνικής θάλασσας όπου τελευταία έχουν δημιουργηθεί αρκετά θέματα. Δεν έχει κλιμακωθεί η σύγκρουση, αλλά παρόλα αυτά ζητάμε από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην κλιμακώνουν την στρατιωτική ένταση, αλλά μέσω διαπραγματεύσεων να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Επίσης ανησυχούμε και για τα τεκτενόμενα στην Κορεατική Χερσόνησο, ιδιαίτερα με τα προγράμματα πυρηνικών όπλων της Βόρειας Κορέας. Η Αυστραλία λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουν να είναι ικανοί εταίροι και να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την καλή συνεργασία τους. Η συμφωνία πλαίσιο που θα πρέπει να υπογραφεί πριν το τέλος του χρόνου καλύπτει όλους τους τομείς συνεργασίας. Η συμφωνία αυτή θα προωθήσει την ευημερία και την ε, ηρεμία θα έλεγα σε όλες τις περιοχές μας και στην Ευρώπη και στη δική μας περιοχή και μας επιτρέπει να ασχοληθούμε καλύτερα με θέματα όπως η διεθνής βοήθεια για την αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, η έρευνα, η καινοτομία, η εκπαίδευση, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα προβλήματα τα μεταναστευτικά κτλ. Επίσης υπάρχει και το φόρουμ το οποίο θα ξεκινήσουμε αργότερα σήμερα μαζί με την κυρία Μόγκερίνη. έτσι ώστε οι άνθρωποι με ηγετικές θέσεις θα μπορέσουν να έλθουν σε επαφή από τις δύο περιοχές και να συζητήσουν από κοινού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η σχέση μας ε, τα τελευταία αυτά χρόνια που έχουμε διπλωματικές σχέσεις είναι μια πολύ παραγωγική <laughs> σχέση. Πρέπει να διευρύνουμε την εταιρική σχέση και με την εμπορική συμφωνία που πρέπει να υπογράψουμε. Εμείς και εσείς σίγουρα έχουμε να ωφεληθούμε από την συμφωνία αυτή θα είναι μια εταιρική συμφωνία η οποία αναβασίζεται σε συμπληρωματικούς ρόλους και σε επίπεδο εμπορικό και εδώ ο Στίβ Τσόμπο θα σας τα πει καλύτερα και αναλυτικότερα. Εμείς είμαστε καλά συνδεδεμένοι με τις αναπτυσσόμενες ραχδαία αγορές της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες για την προώθηση της ειρηνικής συνεργασίας στην περιοχή αυτή, κάτι το οποίο ελπίζουμε ότι θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια. Για το Brexit θα ήθελα να ζητήσω από τους Ευρωπαίους να μην το δουν σαν κάτι το οποίο ε, δείχνει ότι είναι κάτι το παρακμιακό. Όχι, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι υπερήφανη για αυτά τα οποία έχει πετύχει στον τομέα και τον οικονομικό και της διατήρησης της ειρήνης θα πρέπει να συνεχίσει την τεράστια προσπάθεια που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αυστραλία ακόμα και μετά το Brexit σε καμία περίπτωση δεν θα μειώσει την προσπάθεια συνεργασίας. Η συνεργασία όλων αυτών των ελεύθερων δημοκρατιών που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα εξελίσσεται μεν, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσει κυρίως τη μακροβιότητά της. <coughs> Euh, Monsieur le Président. Euh, ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα από πλευρά Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου να χαιρετήσω του ε, προσκεκλημένου μα, ε, του δύο υπουργού από την Αυστραλία. Μα τιμούν με τη σημερινή του παρουσία και απευθύνω ένα χαιρετισμό και προ ολόκληρη την αντιπροσωπεία που του συνοδεύει. Υπουργή, κάνουμε μία ανταλλαγή στα πλαίσια ενός ε, περίπλοκου διεθνούς πλαισίου, όπως προανέφερε ο πρόεδρος ε, Μπρόκ. Το διεθνές ε, εμπόριο και οι συνθήκες που ισχύουν αμφισβητούνται όλο ένα και περισσότερο. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τις εργασίες μας, ούτως ώστε οι μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές να είναι υποφελείς για όλους, σε ένα πνεύμα αμοιβαιότητας, και αμοιβαίου ωφέλους, ούτως ώστε να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και στην ε, δημιουργία θέσεων εργασία ε, Η Ένωση και η Αυστραλία ε, φαίνεται να έχουν κοινέ προκλήσεις και κοινέ ευκαιρίες. Η γεωγραφική απόσταση που μας χωρίζει δεν θα πρέπει να μας εμποδίσει από το να υποστηρίξουμε τι κοινέ μα αξίες. Από πλευράς Επιτροπή ΙΝΤΑ θέλω να περάσω το εξή βασικό μήνυμα. Η Ένωση και η Αυστραλία θα είναι ισχυρότερες αν μείνουν ενωμένε, ε, κυρίως μέσα από τις εμπορικές μας σχέσεις. Η Ένωση και η Αυστραλία είναι μια θύρα εισόδου μια υπήρου και μιας ε, ε, περιφερειακής δύναμης με υπεύθυνη διαχείριση των σχέσεων της παγκοσμιοποίησης, των παγκοσμιοποιημένων εμπορικών σχέσεων και επενδύσεων θα είμαστε ισχυρότεροι ε, αποδίδουμε έμφαση στην ανάπτυξη των σχέσεών μας, κυρίως η Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου που συνέστησε μια ομάδα παρακολούθησης ειδική για την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Επίσης με ενδιαφέρον παρατηρούμε τη συμμετοχή σας στις πολύπλευρες πολυμερής διαπραγματεύσεις όπως για την ΤΙΖΑ, για τα περιβαλλοντικά αγαθά και Επίσης υποστηρίζουμε την πρόθεσή σας ε, να δεχτείτε ε, και τις κρατικές προμήθειες ε, στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Τέλος, το Κοινοβούλιο το Φεβρουάριο ενέκρινε τη θέση του για την έναρξη των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή μιας διμερούς συμφωνίας και ελπίζω η εντολή να είναι διαθέσιμη σύντομα. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε τον Υπουργό υπεύθυνο για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Ο κ. Τσεβού έχει το λόγο. Well, Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ, κυρία Σαϊφή. Και σας κύριε Πρόεδρε Μπροκ. Μεγάλη χαρά και τιμή για μένα να μπορώ να σας απευθύνω το λόγο σήμερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί σας για το βάθεμα <clears throat> των ε, δεσμών εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ των ανοιχτών, ελευθερωμένων και προηγμένων οικονομιών μας. Είμαστε ως Αυστραλία αποφασισμένοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη για την ταχεία προώθηση των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου και θα συζητήσουμε και με όλους τους ευρωβουλευτές. Μια συμφωνία διμερής ελευθέρου εμπορίου που θα πηγαίνει σε βάθος μεταξύ των οικονομιών μας θα προσφέρει δυνατότητες περισσότερου εμπορίου σε αγαθά και υπηρεσίες και αμοιβέ επενδύσεις. Το ίδιο σημαντικό είναι, διότι και οι δυο είμαστε προηγμένες, και και ε, προηγμένες οικονομίες, θα βάλουμε και το ορόσημο για το τι μπορεί να πετύχουν τέτοιε συμφωνίες, διμερεί συμφωνίε ελευθερών εμπορίου μεταξύ ε, εταίρων με παρόμοια νοοτροπία. Θα προφελεί συνεργασία σε τομείς όπως προδιαγραφές, ρύθμιση, ψηφιακή οικονομία, έρευνα και καινοτομία. Τέτοια συμφωνία, FTA, μεταξύ Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτρέψει να προωθήσουμε το κοινό όραμα που έχουμε για το μέλλον του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος. Ήδη συνεργαζόμαστε σε πολλά στοιχεία του διεθνούς εμπορίου και επενδύσεων. Έχουμε κοινό συμφέρον για να προωθήσουμε ένα ισχυρό πολυμερές σύστημα εμπορίου που αναβασίζεται σε κανόνες. Συνεργαζόμαστε σε έναν αριθμό πλειονομερών πρωτοβουλειών συμφωνίες TSA, δηλαδή συμφωνίες και για την εμπορία υπηρεσιών, που είναι σημαντικές για την ε, μελλοντική υγεία, υγεία της παγκόσμιας οικονομίας. Μια συμφωνία μεταξύ Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ενισχύσει τους ε, υπάρχοντες ήδη οικονομικούς δεσμούς. Παρόλο που δεν εμφανίζεται τόσο πολύ στα επίσημα στατιστικά στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός προορισμός και για τις αλλοδαπές επενδύσεις από την Αυστραλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ο μεγαλύτερος εταίρος της επενδύσεις της Αυστραλίας. Κάποιες από τις επενδύσεις αυτές που έρχονται από την Ευρώπη προς την Αυστραλία δηλαδή χρησιμοποιούν την Αυστραλία ως εφαλτήριο για να διασυνδεθούν με τις μεγάλες αγορές της Ασίας. Οι δασμοί μεταξύ Αυστραλία και Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σχετικά χαμηλοί κατά μέσον όρο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι τομεί όπου υπάρχει ακόμα υψηλό επίπεδο προστατευτισμού. Είναι σημαντικό μια διμερής συμφωνία να θέσει τους όρους για ανοιχτό, έντιμο και ισοδίκαιο εμπόριο σε τρόφιμα και αγροτικά προϊόντα, ανάλογα και με τα ε, συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Έχει καλό ιστορικό η Αυστραλία διαπραγματεύσεων ε, σε σημαντικές συμφωνίες με άλλους εταίρους σε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ευκαιρία να συζητήσουμε με την Ευρώπη για τα θέματα αυτά. Σήμερα η φήμη της Αυστραλίας για καθαρή αγροτική παραγωγή είναι γνωστή σε ολόκληρη την Ασία. Ωστόσο, ίσως αυτή η καλή φήμη να έχει δημιουργήσει και τον μύθο ότι οι αγροτικές εξαγωγές της Αυστραλίας είναι μεγαλύτερες από, σε όγκο από ό,τι είναι πραγματικά. Στην πραγματικότητα, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Αυστραλία είναι τετραπλάσιες σε αξία από τις Αυστραλιανές και ούτως ή άλλως η Ευρώπη παράγει 10 φορές περισσότερα από ό,τι εμείς. Για τις υπηρεσίες, η Αυστραλία επιδιώκει μέσω των συμφωνιών ελευθέρου εμπορίου να επιτύχει τα, σε βάθος αποτελέσματα. Προσεγγίζουμε τις διαπραγματεύσεις με τον στόχο να απαλείψουμε ή να ελαχιστοποιήσουμε τους φραγμούς σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς και να βελτιώσουμε τη διαφάνεια. Η συμφωνία FTA με την Ευρωπαϊκή Ένωση μας προσφέρει μία ακόμη ευκαιρία για να προωθήσουμε συμφωνίες και υπέρ των επαγγελματιών μας για τις επαγγελματικές άδειες και προσόντα. Αναμένουμε μια FTA η οποία θα είναι αμοιβαία επωφελής. Θα επιτρέψει να διευκολυνθούν οι επενδύσεις και να προσφέρει αυξημένη ασφάλεια στους επενδυτές και βεβαίως με ταυτόχρονη ε, προσοχή στο δημόσιο συμφέρον. Και οι δύο πλευρές έχουν στέρεα και διαφανή νομικά συστήματα. Άλλο θετικό αποτέλεσμα της συνεργασίας με ε, εταίρους με παρόμοια ε, νοοτροπία είναι και στο μέτωπο των νομικών ρυθμίσεων. Μπορούμε μεταξύ ανοιχτών απελευθερωμένων οικονομιών να φτιάξουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα προσφέρει μεγαλύτερη βεβαιότητα και ασφάλεια στις επιχειρήσεις και στις μικρές και μέσες επιχειρήσεις δηλαδή, μειώνοντας ταυτόχρονα την γραφειοκρατία. Απευθυνόμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν παράληψή μου να, να, να μην αναφερθώ ειδικότερα στην πνευματική διοκτησία. Επ' αυτού θέλω να πω το εξή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση του είδους one size fits all. Χρειαζόμαστε μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των δικαιούχων, των χρηστών, του κοινού και του κρατικού, του δημοσίου συμφέροντος. Στις πρόσφατες FTA έχουμε βρει καινοτόμου τρόπου για να αναγνωρίσουμε το ρόλο τη τεχνολογία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στι διαπραγματεύσει μα με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένουμε να καινοτομήσουν ακόμα περισσότερο προς το κοινό μας συμφέρον και για κοινέ προσεγγίσεις, σφυριλατώντας έτσι την ανάπτυξη στην ψηφιακή οικονομία που είναι σημαντική στόχευση για την Αυστραλία στο διεθνές της εμπόριο και βεβαίως και στις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες ελευθερών εμπόριου. Οι τέτοιες διαπραγματεύσεις είναι περίπλοκες και σίγουρα θα θίξουν και κάποια ε, ζητήματα ιδιαίτερης ευαισθησίας. Στην φάση αυτή της οριοθετήσεως ε, του πεδίου εφαρμογής των συμφωνιών είναι καλό να γνωρίζουμε καθαρά τους στόχους μας, τους αμοιβαίους στόχους μας. Είμαστε δεσμευμένοι να προχωρήσουμε ταχαίως στην έλευση των διαπραγματεύσεων. Από την ε, οπτική γωνία της Αυστραλίας είναι σαφές ότι η διμερής FTA είναι μια ιδέα που έχει οριμάσει πλέον. Και είναι σωστό να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση αυτή με προσπάθειες και από τις δύο πλευρές για να δώσουμε ένα θετικό παράδειγμα στο παγκόσμιο σύστημα εμπόριου. Αναμένω με ενδιαφέρον το άνοιγμα του διαλόγου με τους ευρωβουλευτές μέσα σε αυτή την πρωτοβουλία. Και ως ε, Υπουργό Εμπορίου, συμφωνώ με την Υπουργό μας των Εξωτερικών, λέγοντας ότι συμφωνούμε σε πολλά από τα όσα είπε η κυρία Αντιπρόεδρος και αναμένουμε με ενδιαφέρον και ανυπομονησία να συνεργαστούμε μαζί σας για να προωθήσουμε το κοινό συμφέρον και των δύο πλευρών, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αυστραλίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you for statements. I think that... Ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρεμβάσεις σας. Νομίζω μας προσφέρατε υλικό για συζήτηση και ας αρχίσουμε αμέσως με τον ε, συνάδελφό μου Μιχαήλ Γκάλερ. Προσοχή όμως, θα μιλήσω γερμανικά. Ευχαριστώ πολύ και καλώς ήλθατε και εσείς κυρία Υπουργέ και εσείς κύριε Υπουργέ και μου φαίνεται σωστό και καλό που έχουμε έναν μακρινό αλλά ισχυρό εταίρο και για το εξωτερικό εμπόριο έχω να πω ακόμη ότι θα χαρώ πολύ να μπορέσουμε να συνάψουμε μια καλή θετική FTA με την Αυστραλία. Εγώ του άλλου υποστηρίζω και τι άλλε συμφωνίε που βρίσκονται τώρα στην φάση των διαπραγματεύσεων όπω TTIP ή SETA. οποίο έχει κάποιο καλό προϊόν να πωλήσει δεν έχει κανένα λόγο να φοβείται ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός και δεν θα τα καταφέρει. Από την άλλη μεριά υπάρχει και το θέμα του προσφυγικού το ποια πράγματα συγκρίνονται στην πράξη και ποια όχι από αυτά που κάνουμε, θα γνωρίζετε βεβαίως και εσείς ότι και στην Ευρώπη υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι πρέπει να βρούμε κάποια νησιά στη Μεσόγειο και να τα κάνουμε στρατόπεδα προσφύγων. Και εσείς ε, υπάρχουν ορισμένα, ε, κάνετε κάτι τέτοια πράγματα σε νησιά της Παππούα Νέας Γουινέας αλλά ε, βεβαίως έχει αρχίσει να επιλαμβάνει τώρα το συνταγματικό σας δικαστήριο. Θεωρείτε ότι μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να έχει κάποια επιτυχία στην Ευρώπη. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας εμπειρίες για το προσφυγικό. Και για ένα άλλο σύνολο θεμάτων, έχουμε τη συνεργασία στα πλαίσια των ε, ΑΚΕ, χωρών Αφρικής, Καραβικής, Ειρηνικού και Συμφωνία Κοτονού. Εσείς έχετε επίσης ε, εμπορικές ε, ε, επαφές με τα νησιά της Καραϊβικής. Βλέπετε τη δυνατότητα από την πλευρά σας, για παράδειγμα σε τομείς όπως η συνεργασία στην ανάπτυξη ή και στην ασφάλεια. Υπάρχουν εκεί, υπάρχουν εκεί πράγματα που θα θέλατε να να, δείτε, να συμβαίνουν. Ευχαριστώ. Sorry, I hear you, um, συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Θέλω να... Α, ένα λεπτό να σας καλωσορίσω πρώτα. Ε, απευθύνω τα ερωτήματά μου στον Υπουργό Εμπορίου. Περισσότερο. Με ενδιαφέρουν αυτά που είπατε για τις επενδύσεις και φυσικά από την Αυστραλία προς την Ευρώπη και αντίστροφα υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες επενδυτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνεται προς μια νέα μορφή ένα νέο σύστημα επενδυτικό ε, κυρίως ως προς το ISTS για την διευθέτηση διαφορών. Ε, θα μπορούσατε ενδεχομένως, λαμβάνοντας αυτό υπόψη, να μας πείτε αν ε, θα μπορούσε η Αυστραλία να προσχωρήσει ένα τέτοιο νέο διεθνές σύστημα ή θα έπρεπε να προβληθεί κάτι σε μια διμερή συμφωνία. Για το Brexit, με θα, θα μου πείτε ότι δεν διαπραγματεύεστε με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παρόλα αυτά ήθελα στα πλαίσια ε, των σχέσεων σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και των διμερών σας σχέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, στο μέτρο που ακόμη είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται λοιπόν να διαπραγματεύεστε με μια μικρότερη εντότητα ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω, θα μου πείτε, δεν υπάρχουν επίσημες διαπραγματεύσεις. Ε, και τις ονομάζετε συζητήσεις και όχι διαπραγματεύσεις αυτές τις επαφές που έχουμε. Πώς γίνεται εκ παραλλήλου ε, να υπάρχουν αυτές οι διαδικασίες. Εγώ είμαι Βρετανός και ανησυχούμε θα χρησιμοποιήσετε ως αντάλλαγμα το Ηνωμένο Βασίλειο στις διαπραγματεύσεις. Ε, να πείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίστε μας υπόσχεται το Ηνωμένο Βασίλειο αυτό, εσείς δεν μας το υπόσχεστε και αν το χρησιμοποιήσετε ως διαπραγματευτικό όπλο. Δεν ικανοποιητικό. Ως ε, Βρετανός βουλευτής ε, θα ήθελα να σε απευθύνω αυτή την έκκληση να μην κάνετε διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο με την Ένωση. Τέλος. Κίνα. Ε, έπετε για το καθεστώ ε, οικονομία τη αγορά πολύ δύσκολη απόφαση για την Κίνα και είπατε, αναφερθήκατε στου εξαιρετικά στενού ε, δεσμού με την Κίνα. Τη έχετε ήδη χορηγήσει αυτό το καθεστώ. Ε, μπορείτε να μας σχολιάσετε αυτό το ζήτημα ε, από τη δική σας εμπειρία. Πώς αντιλαμβάνεστε αυτό το θέμα της, του καθεστώ της οικονομίας αγοράς. ευχαριστώ, Τάνοκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλωσορίζω θερμά ε, τους Υπουργούς Μπίσοπε και Τσάβο. Ε, άλλος ένας Βρετανός Ευρωβουλευτής που θα εκλείψει σε λίγο. Είμαι από τις τελευταίες των Μαϊκανών. Ε, οι συντηρητικοί του ECR ε, σας καλωσορίζουν στο Κοινοβούλιο. Σίγουρα ε, ο ευρωσκεπτικός τύπος θα αναρωτηθεί τι χάνεται χρόνο τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ υπάρχει πολλά υποσχόμενη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με το Ηνωμένο Βασίλειο και θα ανθίσουν οι εμπορικές σχέσεις. Όπως είπε και ο κύριος Μάρτιν, αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μετά το Brexit φυσικά με τα στοιχεία που έχουμε τώρα βλέπουμε ότι είναι μόνο 2% του εξωτερικού μας εμπορίου ε, ενώ με το υπόλοιπο της Ευρωπαϊκής είναι 45% και 12% με την ΣΥΠΑ. Ας τα βάλουμε όλα σε μια γενικότερη εικόνα. Σίγουρα οι, οι διμερείς σχέσεις μας ε, ενδεχομένως να επιστρέψουν στο χρυσό αιώνα πρωτού πριν την προσχώρησή μας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πάντως, ε, ε, επειδή είμαστε ακόμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια καθόλου τυπικά, εντάξει διαδικασία για τις διαπραγματεύσεις ως προς τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου. Ε, μας μιλάτε για, ε, για τη συνεργασία μας σε, σε, θέματα ασφάλειας, άμυνας, τον αγώνα κατά των τζιχαντιστών. Εδώ και δεκαετίες είσαστε βασικός πάροχος αγαθών στο βιομηχανοποιημένο κόσμο, βασικός παίκτη ε, στον ειρηνικό, νότια, ε, βόρεια Κορέα, νότια συνική θάλασσα. Έχουμε πολλές κοινέ απόψεις. Όμως δεν αναφερθεί στι σε κάτι άλλο. Ε, στις μεταναστευτικές ροές έχετε μακρά εμπειρία ε, για την αποτροπή της ελαθρέας μετανάστευσης. Ε, είναι ζήτημα κλειδί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε πρόβλημα στη Μεσόγειο και στη Βόρεια Αφρική και μεγάλες μεταναστευτικές ροές, ε, παράνομες και νόμιμες εμείς θα είμαστε οι καλύτεροι φίλοι σας ε, ε, μετά τον Brexit, αλλά αυτό που ε, με χαροποίησε είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα υιοθετήσει ένα σύστημα βάση πόντων όπως το, η Αυστραλία μετά το Brexit για όσους θέλουν να μπουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό το ανέφεραν οι επικριτές Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρόνια. Τώρα ε, στην Νοτιοανατολική Ασία δέχεστε πολύ περισσότερους μετανάστες από ό,τι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και επίσης Ευρωπαίους μετανάστες ε, ε από την Ελλάδα και την Ιταλία, 80.000 παραδείγματο χάρη. Ε, πολύ στενέ σχέσεις έχετε με το Ηνωμένο Βασίλειο και με την Ήπειρο γενικότερα και στα πλαίσια των διεθνών σας σχέσεων θα ήθελα να πω ότι η πολιτική ομάδα ECR που εκπροσωπώ εδώ, δεν είναι οι συναδέλφοι εδώ, αλλά μιλάω εξ ονόματός τους, ακόμη και χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την βάθηση των σχέσεών μας και την υλοποίηση μιας συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αυστραλίας. Ευχαριστώ. Señores ministros, Κύριε Υπουργή, καλώς ήλθατε. Έχετε την υποστήριξη και από πλευράς μου και από πλευράς της φιλελεύθερης ομάδας έτσι ώστε να υπογραφεί το ταχύτερο η εμπορική συμφωνία. Θέσω κάποιες ερωτήσεις κυρίως προς την Υπουργό Εξωτερικών. Σχετικά με τα συμφέροντα στη Συνική Θάλασσα της ε, Λαϊκής Κίνας δημιουργεί ένα τεράστιο πολεμικό στόλο μεταξύ των οποίων ναυπηγεί συνεχώς και αεροπλανοφόρα ε, για να εδραιώσει τα συμφέροντά της και να επηρεάσει τα πράγματα ακόμα περισσότερο και στο βόρειο ειρηνικό και στο νότιο ειρηνικό και αυτό δημιουργεί προβλήματα και σε μικρά κράτη όπως οι Μαριάνες και το Παλάου. Έχετε μια ξεκάθαρη ε, άποψη για νησιωτικά κράτη όπως η Παππούα Νέα Γουινέα, το Κυριμπάτι, το Τουβαλού και άλλες χώρες της περιοχής και πόσο επηρεάζονται από την πολιτική της λαϊκής Κίνας. Ποια είναι η άποψή σας επίσης και η προσπάθεια που γίνεται για την διαμόρφωση νέων υποδομών μεταφορών και επικοινωνίας ανάμεσα σε περιοχές της Κεντρικής Ασίας που ευνοούν και αυτές την κινέζικη παρουσία. Εγώ είναι ένας από αυτούς οι οποίοι έχουν υποστηρίξει περισσότερο την άποψη της ε, εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αυστραλία είναι μονόπλευρες η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρηθεί ένα μεγάλο μπλοκ, είναι ο μεγαλύτερος έτσι και αλλιώ εμπορικός εταίρος. Το 59 όμως της 100 του συνόλου των εμπορικών σχέσεων προέρχεται από, την, από το Ηνωμένο Βασίλειο και το 60% των εξαγωγών οδεύουν προς το Ηνωμένο Βασίλειο. European Union. EU e country, I Νομίζω ότι η παρουσία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι σημαντική, αλλά ακριβώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντική για την Αυστραλία, επειδή το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικό για την Αυστραλία. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και σε οικονομικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Πέρα από το εμπόριο, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μια μεγάλη διεθνής ε, ε, θα έλεγα ε, δύναμη η οποία εξακολουθεί να έχει τη δική της αυτονομία. Ο πρόεδρος διακόπτει τον ομιλητή λέγοντας ότι δεν κάνετε ομιλία τώρα για τα ωφέλη του Brexit. Θα πρέπει να συνεχιστούν, λέει ο ομιλητής οι οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσες έχουν απομείνει, και υποστηρίζουμε την ενίσχυση των σχέσεων αυτών. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου διεθνιστή και θέλω η χώρα μου να έχει στενότατες σχέσεις με όλες τις περιοχές του κόσμου. Και πιστεύω ότι η Αυστραλία μπορεί να καταστεί ο πρώτος εμπορικός εταίρος στα πλαίσια της νέας περίοδου. Και θα πρέπει να υπογραφεί σύντομα η συμφωνία εμπορική ανάμεσα στη χώρα μου και την Αυστραλία, όπως και η συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία. Όλα αυτά έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν και στο εσωτερικό της κοινοπολιτείας, Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ειρήνη και την ευημαρία των λαών των περιοχών μας. Θα φύγει η αντιπροσωπεία και πρέπει να έχουμε και χρόνο για να απαντήσουν. Ε, Υπουργή, εδώ είμαι. Ε, χαίρομαι πάρα πολύ που τονίσατε πως... Ε, Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής για τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο περιοχές μας και ένα θέμα το οποίο τίθεται βέβαια και παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον είναι το θέμα των επενδύσεων και της προστασίας των επενδύσεων. Οι εμπορικές σχέσεις που έχουμε μαζί σας και οι εμπορικές σχέσεις που έχουμε και με την Ιαπωνία δεν έχουν άμεση σχέση με αυτά τα οποία λέγουμε για το TTIP ε, πιστεύω ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν, να δημιουργήσουμε ένα διακανονιστικό πλαίσιο που θα βελτιώσει την οικονομική ατμόσφαιρα ε, των σχέσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε Μπροκ και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω, λέει ο κύριος Ντεκάστρο, του συναδέλφους. Είναι μια ευαίσθητη στιγμή στις σχέσεις μας με την Αυστραλία μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών. Η Επιτροπή Γεωργίας, την οποία εκπροσωπώ, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπάρχει μια σκιά την οποία θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση. Στις 11 ε, του προηγούμενου μήνα η Επιτροπή Αντιντάμπινγκ ε, ε, της Αυστραλίας επέβαλε ειδικούς δασμούς στην εξαγωγή ντομάτα σε κονσέρβα, επεξεργασμένης ντομάτας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους λόγους. Εμείς ε, λαμβάνοντας υπόψη το ότι έχουμε προωθήσει το λεγόμενο Green Box στην Γεωργία, υποχρεώνουμε τους γεωργούς μας σε ένα μεγάλο βαθμό να σέβονται το, ε, την, ε, το περιβάλλον και γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στη συνεργασία ανάμεσα στην Αυστραλία και την Ευρώπη. Τακούλα. Ο κύριος Τάκουλα. Ευχαριστώ. Ε, Υπουργέ Μπίσοπ, ε, καλωσορίσατε. Ε, Υπουργέ Τσόβο, καλωσορίσατε στο Κοινοβούλιο, όπως και ο συνάδελφος Ντέβιτ Μάρτιν ανησυχώ. Θέλω ε, να ξέρω ποια άποψη έχετε σε σχέση με τη διερεύνηση των επαφών με το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ακόμη δεν έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, στην Κίνα, στο, στο G20, ε, είπε ε, ο κύριος Ομπάμα στην Τερέζα Μέη ότι η προτεραιότητα τον είπα, είναι συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι με το ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, ποια είναι η δική σας προτεραιότητα, ε, ε, συμφωνία ελευθέρω εμπορίου με την Ένωση ή με το, το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, ως Φιλανδός Ευρωβουλευτής ε, με ενδιαφέρει να ξέρω ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, των κυρώσεων τη Ρωσία για την Αυστραλία. Εσείς υποφέρατε πολύ με τις κυρώσεις τις ρωσικές για τα γαλακτοκομικά. Μπορείτε να κάνετε μια επισκόπηση πώς επί... σας επηρέασαν οι κυρώσεις που έβαλε η Ρωσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλώς ήλθατε και από μένα. Η ε, κυρία Γκράσφαντερ. Σημαντική η εμπορική συμφωνία, όμως ο στόχος της πρέπει να είναι η αύξηση της ευημερία του κοινού, όχι των επιχειρήσεων. Γνωρίζετε ότι εδώ εμείς ασκούμε κριτική σε ορισμένες συμφωνίες όπως ΣΕΤΑ και TTIP ειδικά για θέματα όπως προστασία επενδύσεων, όπως ε, η αηφορία, η βιωσιμότητα δηλαδή της ανάπτυξης, ότι ε, ανησυχούμε ότι μπορεί ορισμένα παραδοσιακά προϊόντα μας να υποστούν βλάβη και ούτω καθεξής. Έχετε υπόψη σας τα στοιχεία αυτά, έτσι ώστε η συμφωνία να καταλήξει τελικά υπέρ του συμφέροντος και των λαών και των δύο πλευρών. Μια παρατήρηση λέει ο κ σχέσεις μας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί στην ε, περίπτωση αυτή το ε, Brexit, το ενδεχόμενο του Brexit. Εγώ θεωρώ αυτονόητο η Αυστραλία θα ε, συνάψει εμπορική συμφωνία και με την Μεγάλη Βρετανία. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρξει κάποια αντιπαράθεση των θεμάτων αυτών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ωστόσο άκουσα του συναδέλφους Μάρτιν και Τανόκ που έβαλαν το Ενωμένο Βασίλειο να περιμένει στη σειρά. Η Υπουργό Εξωτερικών. Τέθηκαν και ορισμένες ερωτήσεις σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών και γι' αυτό θα ξεκινήσω από αυτές. Το θέμα των προσφύγων και οι συγκρίσιμες ή μη συγκρίσιμες εμπειρίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Αυστραλία. Φυσικά και έχουμε τις δικές μας εμπειρίες στη διαχείριση μη ελεγχόμενων ροών που ζητούν άσυλο. Η Αυστραλία είναι μια χώρα η οποία εδρεώθηκε ε, στα θέματα της, στη μετανάστευση. Από όλο τον κόσμο ήρθαν άνθρωποι και κατέστησαν την Αυστραλία τη χώρα τους. Είμαστε μία από τις πιο πολιτισμικές, αν θέλετε, χώρες στον κόσμο. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς έχουμε υποδεχθεί πάρα πολλούς ανθρώπους, 835.000 τους έχει δοθεί άσυλο, ε, τους έχουν δοθεί θεωρήσεις ανθρωπιστικές που τους δίδουν την δυνατότητα εγκατάστασης στην Αυστραλία. 80.000 ε, το χρόνο είναι διαθέσιμες τέτοιες θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους. Έχουμε επίσης δώσει και άλλες 12 θέσεις μόνιμες επανεγκατάστασης για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν από τη σύγκρουση στη Συρία. Γύρω στους 200.000 ανθρώπους ε, υποδεχόμαστε το χρόνο και εδώ και αρκετά χρόνια Δυστυχώς το λαθρεμπόριο ψυχών, το οποίο είναι στα χέρια φυσικά της οργανωμένης εγκληματικότητας, εκμεταλλεύτηκε τους Αυστραλιανούς νόμους και έτσι πολλοί άνθρωποι από το Ιράν, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν και από την υπόλοιπη Μέση Ανατολή προσπάθησαν να έρθουν στην Αυστραλία πληρώνοντας τους ανθρώπους αυτούς πήγαιναν στην Ινδονησία πρώτα από τη χώρα τους ή στην Μαλαισία και μετά τους έβαζαν σε μία αξιόπλοα σκάφη με Ινδονησιακά πληρώματα και έκαναν πολύ δύσκολα μεγάλα ταξίδια. Γύρω στις 50.000 κόσμος προσπάθησε να το κάνει αυτό, μάλλον 15.000 κόσμος. 1.200 έχασαν τη ζωή τους στα ταξίδια αυτά στη θάλασσα και παρά τις προσπάθειες των σωστικών δυνάμεών μας δεν καταφέραμε να σώσουμε όλους αυτούς. Η εργατική ε, κυβέρνηση ήρθε σε μια συμφωνία με την PNG, την Παππούα Νέα Γουινέα, έτσι ώστε να δώσει και η χώρα αυτή δυνατότητες εγκατάστασης και υποδοχής των ανθρώπων αν είναι γνήσιοι πρόσφυγες. Αλλιώς κανονικά θα βοηθήσουμε την χώρα αυτή που είναι στα βόρεια σύνορά μας να βοηθήσουμε στην παλινόστηση ή καλύτερα στην επαναπροώθηση των, προσφυ... των ανθρώπων αυτών. Ε, συνεχίζεται η συμφωνία αυτή, η εφαρμογή της. Το ίδιο συμβαίνει και με την αντίστοιχη συμφωνία με τον Ναουρού. Ε, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να μπαίνουν και να βγαίνουν στις εγκαταστάσεις τις οποίες έχουν, ε, ζουν, αλλά περιμένουν να εξεταστεί η περίπτωσή τους. Η Αυστραλία λοιπόν έχει σαφείς πλέον κανόνες για τη μετανάστευση. Έχουμε καταστρέψει την διαδικασία αυτή που είχε δημιουργηθεί με την παράνομη μετανάστευση. Δεν έχουν υπάρξει από το 2014 και μετά επιτυχείς τέτοιες προσπάθειες σώματεμπορίας σε εισαγωγικά. Συνεχίζουμε την συνεργασία και με άλλες χώρες της περιοχής ε, για επανεγκαταστάσεις με αυτούς οι οποίοι αναγνωρίζονται ως γνήσιοι πρόσφυγες. Ασχολούμεθα επίσης ε, και με τις χώρες οι οποίες, ε, από τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι δεν την χάνουν αναγνώριση του δικαιώματός τους ως πρόσφυγες. Η εμπειρία της Αυστραλίας δεν μπορεί να αντιγραφεί φυσικά από άλλες χώρες. Βρισκόμαστε σε μια ειδική περίπτωση και περιοχή. Είμαστε μια ήπειρος νήσος και ο κόσμος σε μας έρχεται μετά από ταξίδια χιλιάδων χιλιόμετρων είτε με πλοίο είτε με αεροπλάνο δεν είναι το ίδιο πράγμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά και σε εμά προσπαθούν να έρθουν άνθρωποι για να πετύχουν καλύτερε συνθήκε ζωή. Τέθηκε το θέμα επίση της Κίνας και το πόσο ε, εμεί ασχολούμεθα με την περίπτωση του, ανόδου του καθεστώτος της ε, Κίνα, αν θέλετε, στον κόσμο. Ξέρετε ότι έχει μεγάλη οικονομική σημασία η Κίνα. 140 χώρες έχουν σαν πρώτο οικονομικό εταίρο την Κίνα και μεταξύ τους είναι και η Αυστραλία. Είναι η δεύτερη πιο μεγάλη οικονομική δύναμη. Η Κίνα λοιπόν έχει αυξήσει τις στρατιωτικές της ικανότητες. Ε, η ειρηνική ανάπτυξη της Κίνας είναι κάτι το καλοδεχούμενο. Η Κίνα προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή της ε, αυξάνει την σημασία της σε μια περιοχή στην οποία ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένας ρόλος προστασίας μετά από τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί. Η Κίνα έχει πάρα πολλά να προσφέρει στην περιοχή μας πάντως. Η Κίνα βοηθά και στον τομέα της ανάπτυξης και συνεργασίας. Το πνεύμα συνεργασίας το οποίο επιδεικνύει στον Ειρηνικό ωκεανό βοηθώντας τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι κάτι το ιδιαίτερο θετικό. Το θέμα της ε, νότιας συνικής θάλασσας είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή ε, υπάρχουν ε, διεκδικήσεις ανάμεσα σε διάφορες χώρες όπως η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και άλλες πρέπει οι διαφορές αυτές να αντιμετωπιστούν μέσω ειρηνικών διαπραγματεύσεων να αποφευθεί η χρήση όπλων και να αναζητηθεί επίσης και η διεθνής διαιτησία και διαμεσολάβηση όπως το έχουν κάνει οι Φιλιππίνες. Η Κίνα έχει πάρει ορισμένα ατόλ και ορισμένες βραχονισίδες της περιοχής και τα έχει μετατρέψει σε νησιωτικές δομές, τα έχει καταστήσει ε, στρατιωτικές περιοχές και άλλες χώρες το έχουν κάνει αυτό, αλλά η ταχύτητα και το εύρος της κινέζικης προσπάθειας είναι άνευ συγκρίσεως. Οφείλουμε λοιπόν εμείς να εξετάζουμε την κατάσταση αυτή προσεπτικά, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε το δικαίωμά μας, δικαίωμα υπέρπτυσης των διεθνών υδάτων όπως και οι άλλες χώρες της περιοχής και ουσιαστικά να ασκούμε τα δικαιώματα τα οποία μας δίδει το διεθνές δίκαιο. Ζητούμε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε όλες οι χώρες να σέβονται την κυριαρχία των άλλων χωρών, το διεθνές ένομο καθεστώς, τις διεθνείς ρυθμίσεις και τα θέματα της περιοχής πρέπει να επιληθούν με ειρηνικό τρόπο. Και εδώ έρχεται το θέμα της Ρωσίας εμείς είδαμε ποιες είναι οι ρωσικές ενέργειες σε σχέση με την Ουκρανία. Είδαμε επίσης την προσάρτηση της ε, Κρυμαίας, ήταν μια ύβριση στην διεθνή τάξη ε, και την κυριαρχία φυσικά της ίδιας της Ουκρανίας. Και συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλαμε ε, ε, κυρώσεις εμπορικές οικονομικές στην Ρωσία. Δεν έχουμε πολύ σημαντικές οικονομικές σχέσεις με την Ρωσία. Κυρίως εφήγησαν εξαγωγές μας στον τομέα της γεωργίας. Και, και η Ρωσία φυσικά αντέδρασε στο ίδιο επίπεδο. Πιστεύουμε ότι όταν μια χώρα, όταν ένα έθνος με επιθετικό και μονομερή τρόπο ασκεί αυτό που θεωρεί δικαίωμά του και απαρνείται την κυριαρχία μιας άλλης χώρας, χώρες όπως η Αυστραλία και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει σαφώς να αντιδράσουν και να ζητήσουν την εφαρμογή των προτύπων ε, τα οποία εφαρμόζουν και θέλουν να γίνονται σεβαστά. Thank you uh, Υπουργό Εμπορίου. Ευχαριστώ να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις. Βεβαίως στοχεύσατε πολύ στις ερωτήσεις σας και στις επιπτώσεις ε, της Βρετανικής εξόδου. Όπως είπε και ο πρόεδρος σας, δεν θα έπρεπε να έρχονται σε αντιπαράθεση τα πράγματα αυτά. Θα σας πω λίγα γι' αυτό. Πρώτα για τα δικαστήρια, για την δικαστική επίλυση διαφορών σχετικά με τις επενδύσεις ε, για το σύστημα ISTS. Έχουμε διαξαχάγει συζητήσεις με την Σεσίλια Μάλστρομ. Εάν θα είναι μια ρύθμιση ε, διαρκούς χαρακτήρα ή αν θα είναι, αν θα είναι εξειδικευμένη. Εμείς έχουμε δει ότι λειτουργεί καλά το ISDS. Βεβαίως, ε, ευχαρίστως θα ε, εξακολουθήσουμε να ε, εξετάζουμε το ενδεχόμενο εφαρμογή του συστήματος και στα πλαίσια των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά την Κίνα και το καθεστώς οικονομία τη αγορά. Η δική μας εμπειρία ω τώρα υπήρξε θετική. Βέβαια για μας η Κίνα είναι ε, πολύ σημαντικό εταίρο. Ίσως υπάρξουν κάποιες ε, ε, επιπτώσεις στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου. Αλλά πάντω, επαναλαμβάνω, δεν υπήρξαν αρνητικές οι εμπειρίες μας. Για τα δύο μείζωνα θέματα, κυρίως για το Brexit δηλαδή πρώτα, Αυτό βρίσκει μεγάλη απίχυση και στον Αυστραλιανό τύπο και στον Βρετανικό, ότι οι συζητήσει δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ πιο προχωρημένες και πολύ πιο όριμε σε ό,τι αφορά την ε, προσέγγιση μας ε, για μια ε, Free Trade Agreement. Ελπίζω ότι μέχρι τέλο του έτου θα ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση της οριοθέτησης, δηλαδή το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας. Εγώ βλέπω και ελπίζω να υλοποιηθεί αυτό, η συμφωνία δηλαδή, ή μάλλον οι διαπραγματεύσεις να αρχίσουν πριν από οποιαδήποτε κίνηση γίνει ε, απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυστραλία και Ηνωμένο Βασίλειο έχουν βεβαίω μια πάρα πολύ στενή σχέση. Από την άλλη πλευρά είναι μια χθεσινή σχέση. Ε, ενώ εξετάζουμε τη σχέση μας τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση από μια σκοπιά του εμπορίου, Τώρα το Ηνωμένο Βασίλειο εξέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Λιάν Φόξ ο ίδιο θεωρεί ότι δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν να γίνει η Βρετανική έξοδο Και αυτό σημαίνει για μένα τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Υπάρχει μια ομάδα αξιωματούχων μας που εξετάζει το θέμα αυτό. Αλλά είναι πολύ πιο επίσημη η ε, διαβούλευση που γίνεται ήδη αυτή τη στιγμή για την οριοθέτηση του εφαρμογή τη συμφωνία αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να αρχίσουμε τι διαπραγματεύσει με την Ευρώπη ήδη τι αρχέ του επόμενου έτου. Εσεί νομίζω με ρωτήσατε σχετικά με τα μεγέθη των εμπορικών σχέσεων εκτός ε, ε, μεγάλη Βρετανία. Ακόμα και αν εξαιρεθεί λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση ο τρίτο κατά σειράν εταίρο μα. Και σε ό,τι αφορά τι επενδύσει επίση μιλούμε για 500 εκατομμύρια ...500 ε, δισεκατομμύρια δολάρια δηλαδή με, με, το, με τη Μεγάλη Βρετανία και ένα ε, ε, επίσης ε, μεγάλο ποσό με, χωρίς την Μεγάλη Βρετανία. Να μην αναμειγνύουμε τα δύο αυτά, τις δύο αυτές σχέσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα, τα ε, συμφέροντα των καταναλωτών, έρχομαι στη δική σας ερώτηση, έχουμε πολύ υψηλές προδιαγραφές για την προστασία των ε, καταναλωτών στην Αυστραλία και νομίζω σε αυτό ε, ε, συμφωνούμε. Ιδίω ό,τι αφορά τι προδιαγραφέ, εμεί δεν θα επιδιώξουμε καμιά αποδυνάμωση των προδιαγραφών ασφαλεία, ποιότητα κλπ. που είναι και από τι υψηλότερε στον κόσμο και οι δικέ μα. Και έρχομαι εδώ, πρόεδρο Σαϊφή ότι έχουμε τις ίδιες, έχουμε κοινέ αξίες στο θέμα αυτό. Είμαι απόλυτα πεπισμένο ότι θα μπορέσουμε να ε, ενισχύσουμε τα συμφέροντα αυτά και μέσα από τις διαπραγματεύσεις για την FTA. Για τις δραστηριότητες ε, για το πράσινο καλάθι και ιδίω για ε, τομάτες σε κονσέρβες, κονσερβοποιημένες τομάτες. Έχουμε ε, μια επιτροπή η οποία έχει αναλάβει μια μελέτη ανάλυσης για το θέμα των Ιταλικών τοματοπολτών. Έχω, ε, μου έθεσαν το θέμα αυτό, αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες σχετικά με τις δραστηριότητε του πράσινου καλαθιού. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζεται τώρα στην Αυστραλία. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μελέτη αυτή. Είναι σημαντικό όμως αυτό το ανεξάρτητο σώμα που ανέφερα να επανεξετάσει το θέμα. Και αυτό γίνεται τώρα στην χώρα μας. Άλλο θέμα, η αξία των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Αυστραλία και με εξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πολύ υψηλή η αξία των επενδύσεων αυτών. Ε, επιχειρήσεις όπως Φεραίρο, Νεστλέ, φαρμακευτικές βιομηχανίες, BASF και άλλες ε, και πάρα πολύ ισχυροί δεσμοί μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας που σημαίνουν ότι μια ολοκληρωμένη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου θα προσφέρει το πλαίσιο για να αναπτυχθούν έτσι περαιτέρω οι σχέσεις αυτές. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και με την υποστήριξη της Επιτροπής σας και των μελών της στις συνομιλίες και ελπίζω να μας δοθεί το ταχύτερο δυνατό η ευκαιρία να αρχίσουμε τις, επίσημε τις επίσημες διαπραγματεύσεις. Σα ευχαριστώ λοιπόν για την ευκαιρία που δώσατε να συνομιλήσουμε σήμερα το πρωί. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο Πρόκ. Πάντω, εμένα μου θυμήσατε πόσο σημαντικό πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ Αυστραλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι πιο σαφές πλέον για μένα και πόσο σημαντική είναι η συνεργασία και στην προσπάθεια σταθεροποίησης του κόσμου, του, του πλανήτη. Και για το ζήτημα της Συρίας και για το ζήτημα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και νομίζω ότι πρέπει αυτή η Συμφωνία Ελευθέρων Εμπορίου να προωθηθεί το τα, ταχύτερο δυνατό. Σας ευχαριστώ και για τη συνεργασία με την κυρία Μογκερίνη και για την είδηση της, της ομάδας υψηλού επίπεδου για το θέμα της μετανάστευσης Βεβαίως μπορούμε να, μάθουμε, να διδαχθούμε αμοιβαία. Τα προβλήματά σας δεν είναι συγκρίσιμα με τα δικά μας, λόγω αριθμών και λόγω αποστάσεων. Εμείς έχουμε υψηλότερα νούμερα και χαμηλότερες και ε, συντομότερες αποστάσεις. Εσείς έχετε λιγότερα νούμερα, μικρότερα νούμερα και μεγαλύτερες αποστάσεις. Άρα, βεβαίω και οι λύσεις που θα δοθούν δεν μπορούν να είναι απολύτως συγκρίσιμες. Είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να λάβουμε υπόψη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ε, προσήλθατε ενώπιον μας είναι σημαντική τιμή για μας και ίσως η κυρία Σαϊφή θέλει να πει λίγα λόγια ολοκληρώνοντας την συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους Υπουργούς για την παρουσία τους, για τις παρεμβάσεις τους και για το διεθνές εμπόριο. Ε, Είδατε, Υπουργέ Τσιόμπο, πόσο μεγάλο ενδιαφέρον έχουν οι συνάδελφοι για τι ε, επερχόμενε διαπραγματεύσει. Ε, με τα χαρά να σα υποδεχτούμε και πάλι στο Κοινοβούλιο, αυτή τη φορά στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου, για να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε. Μπρόκ, ευχαριστώ. Thank you. go to the mm-hmm.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 Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα. Θα έχουμε την δυνατότητα να ακούσουμε τον κύριο Φρανκ Μπρένερ. Είναι Γενικός Διευθυντής του Aerocontrol και θα μας μιλήσει για την αεροπορική ασφαλεία σε περιοχές ε, συγκρούσεων είναι μια διακυβερνητική διεθνής οργάνωση υπεύθυνη για τη διαχείριση των αερίων μεταφορών, των εναερίων μεταφορών. Ε, υπάρχουν εκατομμύρια πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν ουσιαστικά τις υπηρεσίες της σε ημερήσια βάση. Αυξάνεται συνεχώς ε, ο όγκος των αερομεταφορών στην Ευρώπη πλέον και γίνεται αξιολόγηση των κινδύνων σε συνεργασία με άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως η ΙΚΑΟ. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποιες είναι οι πρώτες ιδέες, τα πρώτα αν θέλετε συμπεράσματα των επαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της αξιολόγησης των κινδύνων και της ανταλλαγής πληροφοριών για την αντιμετώπιση των διεθνών κρίσεων. Συνειδητοποιούμε τις δυσκολίες και τις αντιστάσεις οι οποίες συναντώνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, ε, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτών. Πάντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύουμε ότι το Eurocontrol βοηθά, συνεισφέρει στην δημιουργία ενός ασφαλούς οργανωμένου συστήματος αερομεταφορών και στην Ένωση και στις γειτονικές χώρες. Έχετε το λόγο κύριε Μπρένερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να πάρω το λόγο μπροστά σας σήμερα και να σας ε, ενημερώσω για το πού βρισκόμαστε στο Eurocontrol σε σχέση με την ασφάλεια των ε, ε, μεταφορών. Και αναφερθήκατε και στο θέμα των περιοχών συγκρούσεων. Σας δείχνω εδώ ένα γράφημα για την εξέλιξη της μεσαίας τάξης ε, και το πώς αλλάζει τα τελευταία χρόνια. Over Βλέπετε ότι υπάρχει μια αλλαγή στις συμπεριφορές σε όλο τον κόσμο. Στο παρελθόν η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν ε, το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών μεσαίας τάξης αν θέλετε σε όλο τον κόσμο ενώ τώρα βλέπουμε χώρες κυρίως στην Αφρική, στην Ινδία δηλαδή, αλλά και στην Αφρική που αυξάνεται ε, με πολύ γρήγορο ρυθμό η μεσαία αυτή τάξη και αυτό επηρεάζει φυσικά τα πράγματα και στην Ευρώπη στον τομέα των αερομεταφορών και ε, στην συνδεσιμότητα την οποία επιθυμούμε όλοι μέσω των αερομεταφορών αυτών. Οι αλλαγές αυτές δεν είναι κάτι το οποίο μας προκαλεί έκπληξη. Ε, στην ουσία αντικατοπτρίζονται και στις προβλέψεις των αεροπορικών ροών στις αερομεταφορές στο μέλλον. Αυτή η διαφάνεια δείχνει το πόσο το 2010 ήταν οι αερομεταφορές, σε ποιο σημείο ήταν σε όλο τον κόσμο, το 16% του συνόλου σε επίπεδο εισοδή, μάλλον α, κόστους ανά χιλιόμετρο ανά επιβάτη ήταν το Ευρώπη το 16% λοιπόν. Αυτό άλλαξε και θα αλλάξει ακόμα περισσότερο προς το 2036. Το ποσοστό το ευρωπαϊκό θα πέσει από το 16% στο 11%. Όχι γιατί θα μειωθεί ε, η κίνηση στην Ευρώπη, αντίθετα η κίνηση θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αλλά δεν αυξάνεται τόσο γρήγορα όσο αυξάνεται η κίνηση των επιβατών μέσω αεροπλάνων στον υπόλοιπο κόσμο. Και γι' αυτό ακριβώς σε επίπεδο ποσοστού η Ευρώπη κατεβαίνει αν θέλετε. Στα πλαίσια των 41 μελών ε, του Aerocontrol έχουμε 10 εκατομμύρια πτήσεις κατέτος και ε, το 2036 θα φτάσουμε τα 14 εκατομμύρια ή και τα 15 εκατομμύρια. Υπάρχει λοιπόν τεράστια αύξηση, αλλά παρόλα αυτά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο η αύξηση αυτή είναι μικρή, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ασίας, της Ινδίας και ειδικότερα της Κίνας. Αυτό έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις σε τομείς όπως η ασφάλεια των κινήσεων των αεροσκαφών, και της ε, επικοινωνίας της Ευρώπης με τις χώρες αυτές. Είναι μια ευκαιρία φυσικά και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, γιατί αυτές οι ταχύτατα αναπτυσσόμενες περιοχές έχουν ανάγκη την τεχνογνωσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι προορισμένη αν θέλετε από τη φύση της η Ευρώπη να στηρίξει τις περιοχές αυτές σε επίπεδο τεχνολογίας στον τομέα αναφέρομαι ε, της προστασίας της ασφάλειας στις αερομεταφορές μέσω και της Συμφωνίας Ενιαίας ε, Κάλυψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, στον τομέα της διαχείρισης του εναερίου χώρου ξέρουμε ότι θα υπάρχει αύξηση της δραστηριότητάς μας κατά 25 με 29%. Αυξάνονται επίσης οι πτήσεις χωρίς ενδιάμεσο σταθμό από την Κίνα και την Ασία γενικά προς την Ευρώπη. Βλέπουμε ότι τώρα κυκλοφορούν νέα αεροσκάφη, τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν για πάρα, έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια, εν ακτίνα δράσης να το πω, και ε, βλέπουμε ότι αυτό έχει συνέπειες στα λεγόμενα hubs, στα κέντρα δηλαδή όπου συναντώνται οι πτήσεις και με μικρά αεροσκάφη τώρα συνδέονται ε, πόλεις ε, μεταξύ τους οι οποίες ε, χαρακτηρίζονται ως μικρές πόλεις και πολλές από τις πόλεις αυτές στην Ασία δεν τις γνωρίζουμε καν, αλλά έχουν απευθείας πτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα έχουν ακόμα περισσότερες στο μέλλον απαιτείται σωστή ανταλλαγή απόψεων, ε, ε, ε, στοιχείων μάλλον και πληροφοριών στην Ευρώπη. Το Eurocontrol λοιπόν καλύπτει όχι μόνο τις 28 χώρες, αλλά όπως είπα έχει 41 μέλη συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα έχουμε επικοινωνία με τις περιοχές μεγάλης ανάπτυξης όπως η Λατινική Αμερική η Βραζιλία, τα Ενωμένα Αραβικά Εμμυράτα που είναι μια τεράστια επιχειρηματικά προσπάθεια στον τομέα των αερομεταφορών, αλλά και η Κίνα, η Ινδία και επικοινωνούμε με τις χώρες αυτές και τις κυβερνήσεις τους και τις υπηρεσίες τους έτσι ώστε να συλλέγουμε τα στοιχεία τα οποία απαιτείται να έχουμε. Και το ΙΚΑΟ θεωρεί ότι το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει είναι ένα σύστημα παγκόσμιου ελέγχου των ροών των αεροπορικών. Εμείς ε, λειτουργούμε στα πλαίσια της συνθήκης την οποία πρώτη υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ουρανού αν θέλετε, αλλά ε, όχι μόνο για τις 28 χώρες, αλλά τις 41 χώρες ε, στις οποίες περιλαμβάνεται η Γεωργία και η Αρμενία. Κάναμε συμφωνία και με δύο νέες χώρες, το Βασίλειο του Μαρόκου και το Ισραήλ. Αυτό ε, είναι συμβατό με την ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασίας με την γειτονία και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών μεσογειακού τύπου συμφωνιών, έτσι ώστε και η αγορά η αεροπορική των χωρών αυτών να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς περιορισμούς στην πρόσβαση και στα δικαιώματα πτήσης ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει περαιτέρω επιβατικές και α, τουριστικές μετακινήσεις και αυτό ελπίζουμε θα βοηθήσει γενικότερα στην καλύτερη συνδεσιμότητα σε εισαγωγικά των χωρών μας με αυτές τις χώρες και στη μείωση του κόστους των εισιτηρίων. Η συνεργασία λοιπόν αυτή με το Μαρόκο και το Ισραήλ θα επιτρέψει την ανταλλαγή στοιχείων. Ε, είναι κοντά στην οικογένειά μας οι χώρες αυτές, τα συμμετέχουν πλέον σε όλες τις δραστηριότητες του Aerocontrol είναι σημαντικό γιατί όπως και οι υπόλοιπες χώρες μέλη του Eurocontrol που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβονται τους κανόνες της Συμφωνίας Ευρωπαϊκός Ουρανός. Έτσι θα υπάρξει ένα ομοιογενές πλαίσιο λειτουργίας των ροών ε, των αεροπορικών κινήσεων. Εμείς πιστεύουμε ότι οι χώρες αυτές θα πρέπει να δεχθούν την Συμφωνία Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός και να την εφαρμόσουν πλήρως. Με την ανάπτυξη αυτή μπορούμε να δούμε τώρα ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουμε και έρχομαι στο θέμα των περιοχών σειράξεων. Μετά από την καταστροφή της, ε, που συνέβη στην πτήση Άμστερνταμ Κουάλα Λουμπούρ εμείς ε, ενημερώσαμε όλους τους αερομεταφορείς και τους ευρωπαϊκούς και τους ξένους αερομεταφορείς για τις διαδικασίες ε, στα πλαίσια του προγραμματισμού των πτήσεων υπογραμμίζοντας τους κινδύνους τους οποίους αναφέρουν οι χώρες. Υπάρχει μια χώρα, υπάρχει, μπορεί να υπάρχει θεωρητικά μια χώρα η οποία σημειώνει ότι υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κίνδυνος, ίσως όμως και άλλες χώρες, δεύτερες ή τρίτες χώρες, δημοσιεύουν στοιχεία κινδύνου υψηλού για άλλες περιοχές ή για άλλες χώρες. Αυτό είναι θα έλεγα μια πλατφόρμα η οποία ενημερώνεται συνεχώς σε ζωντανό χρόνο, σε πραγματικό χρόνο ε, και έτσι οι αερομεταφορείς είναι σε θέση να προγραμματίζουν τις πτήσεις τους. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο απευθύνεται μόνο σε ευρωπαϊκούς αερομεταφορείς, αλλά σε όλους τους ε, αερομεταφορείς στον κόσμο. Η πλατφόρμα αυτή είναι προστατευμένη, ε, μπορεί να έχουν πρόσβαση σε αυτήν αυτοί που έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση δηλαδή τα κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΆΣΑ και οι αερομεταφορείς. Ενημερώνεται συνεχώς το site αυτό, είναι ε, θα έλεγα κάτι το θετικό. Αυτό δείχνει όμως και τα προβλήματα που έχουμε στην Ευρώπη με όλο και περισσότερες προειδοποιήσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Η παρατήρηση αυτών των ε, εστιών αν θέλετε ε, συγκρούσεων δημιουργεί κάποια προβλήματα στην σύνδεσή μας σε επίπεδο αερομεταφορών με την Ασία. Διότι οι πτήσεις αναγκαστικά πηγαίνουν από άλλες περιοχές, ε, μειώνεται δηλαδή η δυνατότητα επιλογής δρομολογίων και στην ουσία η υπέρπτυση των περιοχών που βλέπετε στο χάρτη ε, ουσιαστικά απαγορεύεται ή δεν είναι διαθέσιμη στην πραγματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να καταστήσουμε σαν διαχειριστές του δικτύου εύκολη την χρήση και την εκμετάλλευση των αερομεταφορών λειτουργούμε σαν συγκεντρωτικό αν θέλετε σημείο στο οποίο συλλέγονται οι πληροφορίες. Ε, δεν είμαστε η ΆΣΑ. Η ΆΣΑ είναι διακανονιστικό όργανο η οποία ορίζει τους κανόνες, ε, αποφασίζει και ε, ενημερώνει το αεροκοντρόλ, ελέγχει την λειτουργία του αεροκοντρόλ και ελέγχει και τη λειτουργία της πλατφόρμας ενημέρωσης για τις ζώνες κρίσης. Έχουμε ένα μείζωνα ρόλο να παίξουμε λοιπόν σε περιπτώσεις κρίσεων. Εμείς είμαστε το κεντρικό σημείο συλλογής αλλά και διάδοσης της ενημέρωσης. Αυτά μπορεί να είναι συγκρούσει σε τεχνικό επίπεδο, μπορεί να είναι τεχνικά προβλήματα σε τεχνικό επίπεδο που δεν έχουν πολύ μεγάλη δημοσιότητα, τύχη μεγάλης δημοσιότητας. Έχουμε κρίσεις σημαντικές όπως η έκρηξη του ηφαιστείου ε, στην Ισλανδία με την τεράστια συγκέντρωση ηφαιστιακής τάχτης. Ε, είχαν δημιουργηθεί προβλήματα επίσης ε, όπως με τις τρομοκρατικές ενέργειες της Βρυξέλλες όπου τεράστιες ροές έπρεπε να οδηγηθούν σε, άλλα, σε άλλους αερολιμένες γιατί έπρεπε να κλείσει το αεροδρόμιο των Βρυξελών για λόγους ασφαλείας. Όλα αυτά είναι σενάρια κρίσης άμεσα αντιμετωπίσιμα από πλευράς των διεθνών οργανισμών μεταξύ των οποίων και του δικού μας. Ανταλλάξαμε επίσης ε, με ε, τους συνεργάτες μας ε, στοιχεία ευαίσθητα και με χώρες της Ασίας. Ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Aerocontrol να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο όπου συγκεντρώνονται όλα τα δεδομένα των μετακινήσεων των αεροσκαφών. Είναι ένα δίκτυο το οποίο προστατεύεται σε επίπεδο ε, προστασίας ακριβώς των δικτύων, ασφάλειας των δικτύων. Κανένας δεν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ε, στα δίκτυα αυτά. Αποτρέπονται οι επιθέσεις σε ηλεκτρονικό και πληροφορικό επίπεδο. Αυτό λοιπόν αντικατοπτρίζει τις δραστηριότητες ε, τις οποίες έχει αναλάβει ε, το αεροκοντρόλ έτσι ώστε η πτήση σήμερα να είναι ασφαλής. Ε, έχουμε επίσης και την δυνατότητα χρήσης του εναέριου χώρου και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο στρατιωτικό. Δίδουμε προτεραιότητες στον στρατιωτικό τομέα, αν χρειάζεται αυτό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ταυτόχρονα οι ροές προς τις ασιατικές χώρες δεν θα πρέπει να παρεμποδίζονται, διασφαλίσουμε το ανεμπόδιστο των πτήσεων και της ε, ε, αύξησης των πτήσεων αυτών προς την Ασία κυρίως και μάλιστα ε, λειτουργούμε και προληπτικά. Πριν ξεκινήσει μια πτήση γνωρίζουμε το δρομολόγιο, τα ωράρια κτλ. Είναι επιτυχέστατος ο τρόπος λειτουργίας πρέπει να πούμε του Eurocontrol. Είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε τη δραστηριότητά μας η οποία προβλέπεται από τις συμφωνίες μέχρι το 2019 Πρέπει να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η οποία όταν συνετάχθη δεν ήταν τόσο αναλυτική όσο απαιτείται σήμερα να είναι και να καλύπτονται και οι τεχνικές απαιτήσεις αλλά και να διασφαλίζεται η πρόθεση των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης στον κόσμο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα ποιοι συνάδελφοι θέλουν το λόγο. Και ο Γκάλα πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Μπρένερ για την ευρεία επισκόπηση και την εξήγηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε ιδίω σε ζώνες συγκρούσεων που αρχίζουν και πληθαίνουν γύρω μας και που επηρεάζουν βεβαίως τους αεροδιαδρόμους και βεβαίως και τις ικανότητες υπερπτήσεως. Πρόσεξα κιόλας σε πτήσει προς την Μεσημβρινή Αφρική ότι παλαιότερα πετούσαμε πάνω από την Λιβύη, τώρα πηγαίνουμε δυτικότερα πάνω από την Αλγερία. Είναι και ασφαλέστερο ίσως να περάσει κανεί, να περάσει το αεροπλάνο δηλαδή πάνω από Τσάντ και Νίγηρα. Μιλήσατε για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση, που είναι ωστόσο μέλη τη Ευρωκοντρόλ όπως Κάφκασο, αλλά και από την άλλη μεριά το Μαρόκο. με χώρες όπως Αργερία, την Ισία, Αίγυπτος. Υπάρχουν ακόμα κάποιες διαπραγματεύσεις που πρέπει να γίνουν. Για τη Λιβύη δεν μιλώ ακόμη. Δεν είναι καν λειτουργικό κράτος ακόμη. Σχεδιάζεται κάτι. Και ποιες είναι οι επιπτώσεις ό,τι αφορά την ε, μεταφορά δεδομένων. Το Ισραήλ βεβαίως είναι απόλυτα εξοπλισμένο, γνωρίζουν πάρα πολλά και μπορούν ίσως να μας βοηθήσουν προκειμένου έτσι ώστε να αναγνωρίζουμε έγκαιρα ενδεχόμενους κινδύνους αλλά με χώρες όπως το Μαρόκο με το οποίο συνδεόμαστε και στο μέλλον ίσως στην Τινησία αυτές οι χώρες αναμένουν μάλλον από εμάς να βοηθήσουμε τι μπορούμε να τους προσφέρουμε εμείς ως πληροφορίες ασφαλείας Ευχαριστώ κύριε Γκάρε. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωκοντρόλ παρόλο που προκαλεί σύγχυση σε κάποιους ε, εκτός Ένωσης δεν είναι θεσμικό όργανο της Ένωσης και τα μέλη της αριθμούν περισσότερα από τα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης. Μετά από την απόφαση περί Brexit θα χρειαστεί κάποιες ειδικέ αλλαγές ή διαπραγματεύσεις για την Βρετανία ή θα συνεχίσει η Μεγάλη Βρετανία να παραμένει μέλος Ευρωκοντρόλ ανεπηρέαστη ως πλήρες μέλος χωρίς να χρειαστεί να προκληθούν ιδιαίτερες αλλαγές ή συστάσεις. Ο κ. Λόπεθ Ιστούριθ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Είναι μια καλή ευκαιρία σαν πολύ συχνή χρήστη των αερομεταφορών. I και νομίζω ότι πολλοί το ζουν καθημερινά. Δεν θα κάνω εξαίρεση, απλώ θέλω να εκφράσω το σκεπτικισμό μου σε σχέση με του ελέγχου που γίνονται στη Γαλλία. Είναι γνωστό ο εκβιασμό που τον κάνουν κάθε Χριστούγεννα, κάθε καλοκαίρι. Αλλά ξέρω δεν φταίτε εσεί. Δεύτερον, μιλήσατε για τι εμπόλεμε ζώνε και μα δείξατε του χάρτε που έχουν ε, για να προγραμματίσουν τι διαδρομέ και τι πτήσει οι ειδικοί. Θέλω να ρωτήσω το εξή. Μήπω ε, ε, και οι χρήστε να ενημερώνονται άμα είναι να, χρησιμο... να πετάξουν με μια πτήση για να ξέρουν αν πρέπει να την πάρουν ή όχι. 90% των χρηστών ε, με το μαλαισιανό αεροσκάφο δεν ήξεραν κατά πάσα πιθανότητα ότι θα διέρχονταν από ε, επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη. Ε, λοιπόν, καταλαβαίνω ότι για μέτρα ασφαλεία, από πλευρά μέτρων ασφαλεία δεν μπορείτε να τα κοινοποιείτε αυτά. Όμω ε, θέλω να ρωτήσω, δεν πρέπει να ενημερώνονται και οι επιβάτε όταν πρόκειται, πρόκειται η πτήση του να περάσει από τέτοια επικίνδυνη ζώνη. Κύριε Μπρένερ, πολύ χαίρομαι για την ανταλλαγή απόψεων. Όχι μόνο ως Ευρωβουλευτής, αλλά και ως επιβάτης, αλλά και πιλότος. Αναψυχής. Ε, ο, ο, Ευρωπαϊκός Ουρανό είναι πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό πρόγραμμα. Δεν έχει τύχει τις ίδιες προβολές όπως άλλα προγράμματα. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρώπης, όχι μόνο από πλευράς ασφάλειας, αλλά και για άλλους λόγους. Και αυτό το πρόγραμμα Νέος Ευρωπαϊκός Ουρανό προϋποθέτει ότι θα υιοθετήσουμε και ε, ε, μια προσέγγιση στρατηγικού χαρακτήρα, ώστε να είναι βιώσιμη η δράση που αναλαμβάνουμε. Λοιπόν, ε, οι τομεακές στρατηγικές Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να συμπτυχθούν σε μια σφαιρική προσέγγιση που θα εστιάζει όσο επί το πλήθον στην ασφάλεια αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Δύο ερωτήσεις έχω για σας. Ποιο είναι το όραμά σας, αν μπορείτε να σχολιάσετε το θέμα του ε, ε, νέου ευρωπαϊκού ουρανού σε μια δεκαετία. Τι προβλέπετε να συμβεί. Και δεύτερη ερώτηση, με την ιδιότητα του επιβάτη στο Στρασβούργο, ξέρετε εδώ και δύο χρόνια έχουμε την πτήση, αλλά υπάρχουν προβλήματα γιατί είναι ασύμβατα δύο τεχνικά συστήματα. Αυτή που παίρνουν αεροπλάνο από στρασβού ξέρουν πόσο ε, πόση σημασία έχει αυτό για να γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα συστήματα Air France και Lufthansa. Ο κύριος Επιτήδιος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπρέρ που μας ε, είπε αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα και μας έδωσε με αυτό τρόπο να καταλάβουμε πώς ακριβώς λειτουργεί το Eurocontrol. Θα ήθελα να του κάνω μια ερώτηση η οποία αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο ε, επιτυχάνεται η ασφάλεια των πτήσεων σε περιοχές που διεξάγονται πολεμικές επιχειρήσεις. Υπάρχει κάποια συνεργασία με τις δυνάμεις οι οποίες ενεργούν εκεί και κατά δεύτερο λόγο πώς είναι δυνατόν να αποφευθεί μία περιοχή στην οποία δεν διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις, αλλά υπάρχει δυνατότητα κάποια τρομοκρατική οργάνωση να μπορεί να παρέμβει και να απειλήσει την ασφάλεια των επιβατών σε αυτή την περιοχή. Ευχαριστώ. Solo es el tiempo de las respuestas para el señor Brenner, cuando usted quiera. Κύριε Μπρένερ, ήρθε η ώρα των απαντήσεων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. για τις ερωτήσεις Θα προσπαθήσω να σπάρω πάρω με τη σειρά, όπως εσείς θέσατε. Κύριε Γκάλερ, αναφερθήκατε στον ε, στην, ε, στον επαναπρογραμματισμό των διαδρομών για, παράκαμψη των ε, εμπόλεμων ζωνών. Βλέπετε από το χάρτη ότι ε, η Λιβύη για τις υπερπτήσεις δεν είναι η ασφαλέστερη χώρα και αυτή είναι η απόκριση πολλών κρατών και οι αερομεταφορείς το λαμβάνουν υπόψη ως Eurocontrol τους δίνουμε όλες τις διαδρομές, βλέπουμε δηλαδή τα, τις διαδρομές των αερομεταφορέων και κάνουμε έναν έλεγχο ε, για να δούμε αν λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις μας. Εάν όχι, του ενημερώνουμε και πάλι ότι είναι διαθέσιμε οι πληροφορίε Οι αερομεταφορεί δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο και ακολουθούν αυτέ τι συμβουλές για τη Νότια Αφρική, παραδείγματο χάρη παρακάμπτεται η εμπόλεμη ζώνη και ακολουθείται διαδρομή από την ε, Δική Αφρική, πολύ μακρύτερη διαδρομή. Για την ανταλλαγή δεδομένων με διάφορες χώρες, ναι, ναι, δύσκολη ερώτηση σταδιακά θα δούμε τις εξελίξεις με το Βασίλειο του Μαρόκου. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, της συνολικής συμφωνίας, καταλήξαμε στο ότι θα μεταβεί μία ομάδα για το, σε συνεργασία με το RNSP, που είναι η εποπτική αρχή, να δει ποια πρότυπα εφαρμόζονται στο Μαρόκο και αντίστοιχα στον ενίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και ε, συντάσσουμε με την ομάδα εργασία ένα σχέδιο δράση ε, να δούμε ποια υποστήριξη χρειάζεται ούτω ώστε αυτά τα πρότυπα να μετατραπούν σε επίπεδο ε, κατάλληλο για το ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Στην συνεργασία λοιπόν εξετάζουμε τα συστήματα που χρησιμοποιούν και το καλό είναι ότι ανοίγουν τις πόρτες. Ε, δυνάμει αυτής της συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τη συμφωνία Euromed σε πολιτικό επίπεδο και σε τεχνικό επίπεδο με την συμφωνία Eurocontrol που ακολούθησε τη Euromed τη συμφωνία Euromed. Με χαρά και ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν εξελίξεις και όλο και περισσότερα επίπεδα ασφάλειας ε, εγκρίνονται για τον ευρωπαϊκό ουρανό και η ανταλλαγή δεδομένων θα εφαρμοστεί σταδιακά. Αρχίζουμε με μικρά δεδομένα και θα κλιμακώσουμε τη δράση μέχρι δεδομένα από ραντάρ όταν ε, λειτουργούν τα τεχνικά συστήματα και υλοποιηθούν τα μέτρα ασφαλείας. Ε, γίνεται σε βάση need to η ανταλλαγή δεδομένων ε, όταν είναι απαραίτητε οι πληροφορίες. Όταν πάει η πτήση προ το Μαρόκο, τότε δικαιούται αυτά τα δεδομένα το Μαρόκο, αν όχι, όχι. Αυτά προβλέπονται στη συμφωνία και το αντίστροφο ισχύει. Άμα πετάει προς τον Νότο κάποιο από το Μαρόκο, δεν ενδιαφέρει απαραίτητα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, όταν ταξιδεύουν και μπουν στο δικό μα ένα αέριο, μα ενδιαφέρει. Ισραήλ φυσικά είναι σε πολύ προηγμένο τεχνολογικό επίπεδο. Θέλουν ε, να συμβάλλουν ε, στενά στα δικά μας ε, προγράμματα ε, για τη δυναμικότητα. Το μεγάλο αεροδρόμιο του Τελαβίβ έχει περιορισμούς τεχνικούς και πολιτικούς για την πρόσβαση προς τη Μεσόγειο και μόνο, όχι προς άλλες κατευθύνσεις. Τι σημαίνει αυτό, πρέπει να ενορχιστρώνουμε τις ροές με ιδιαίτερα ευφυή τρόπο όταν μπαίνουν ή βγαίνουν από το Ισραήλ Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι η επίπτωση του Brexit ε, για το Ευρωκοντρόλ και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο παρελθόν ήσασταν ε, υπέρμαχος ε, του Eurocontrol που ιδρύθηκε το 1961. Ήταν Βρετανός ο προκάτοχός μου. Και το Ηνωμένο Βασίλειο πάντα κατεδείκνει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ευρωκοντρόλ δεν ε, διαβλέπουμε κάποια ε, μεταστροφή στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το, Brexit, ε, το δημοψήφισμα του Brexit. Ούτε και από πλευράς άλλων διεθνών οργανισμών. Οπότε, οι συζητήσει που έχουμε κάνει με του προς το παρόν δείχνουν τον ενθουσιασμό που υπάρχει να συνεχίσει ο ευρωπαϊκός συντανισμός για να κατοχυρωθούν, να διαφυλαχθούν οι αξίες και τα πρότυπα του ευρωπαϊκού ουρανού στο Ενωμένο Βασίλειο, όπως και σε άλλα μη κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην, Ένωση, ξέρω, έχουμε, ε, στην Ευρώπη έχουμε τα 28 κράτη-μέλη και 13 κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά, ε, αν α, υπάρξει αλλαγή με τον Brexit, θα εφαρμοστεί η κατάλληλη απόφαση, αλλά ε, είναι συμφέρον ε, το Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετάσχει στο, στην δράση του Ευρωκοντρόλ και δεν διαβλέπουμε κάποια, ε, να, να συντρέχει κάποιο λόγο για να αλλάξει η πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου. Λοιπόν, για τι απεργίε. Ναι, εξαιρετικά ενοχλητικό ζήτημα. Μπορούμε εμεί να μπούμε σε εργατικά ζητήματα, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τι κάνουμε, εξετάζουμε τι επιπτώσει των απεργιών. Τρεις τέσσερις είδαμε στη Γαλλία, γιατί αναφέρατε αυτή τη χώρα φέτος. Ένα εκατομμύριο λεπτά καθυστερήσεων για τους επιβάτες, μόνο για φέτος. Και δεν λαμβάνουμε υπόψη ε, τον τεράστιο όγκο πτήσεων που ακυρώθηκαν λόγω της απεργίας. Ε, οι καθυστερήσεις είναι από τις πτήσεις που έγιναν. Είναι πάρα πολύ μεγάλη οικονομική επίπτωση. Πολλοί επιβάτες μένουν εγκλωβισμένοι στα αεροδρόμια. Και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτουμε το ερώτημα δεν πρέπει να υπάρξει μια εναρμόνιση συμφωνής για ελάχιστες υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται ακόμη και όταν υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση. Βάσει εθνικής νομοθεσίας ε, προβλέψε κάποια κράτη μέλη αυτή ελάχιστη υπηρεσία, σε άλλες όχι και πρέπει να ευθυγραμμιστούν αυτές οι εθνικές νομοθεσίες. Εμείς προχωρούμε προς μια σύμφωνη για αποτίμηση της κατάστασης και να δούμε ιδανικά σε νομοθετικό επίπεδο, σε επίπεδο 28 κρατών μελών. Πώ θα διαμορφωνόταν η κατάσταση για να θεσπιστεί μια εναρμονισμένη πρόταση για την ελάχιστη παροχή ελάχιστη καθολική υπηρεσία. Δεν θέλουμε να κουμπίσουμε το θέμα τη απεργία σε καμία περίπτωση. Όμω είναι τόσο μεγάλη η επίπτωση και τόσο ε, διαφορετική ανάλογα με το ποια χώρα μιλάμε, επειδή όλα οργανώνονται εθνικά και δεν υπάρχουν εναρμονισμένε νομοθεσίε, που έχουμε και αυτή την επιδίωξη. Ο στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακρίβεια ε, στις επτήσεις ε, με τις τρεις θέσεις απεργίες δεν είναι εφικτό. Με ένα εκατομμύριο λεπτά καθυστέρηση ακυρώνεται, αναιρείται αυτός ο στόχος. Ε, σε 16 χώρες, επειδή είχαμε θέσει το στόχο σε 0,6 λεπτά αναπτύσσει, πάει, αναιρέθηκε αυτή η πτήση πέρα από αυτές τις απεργίες που σας είπα, γιατί υπάρχει και η καθυστέρηση για διαχείριση εναέρειας κυκλοφορίας. Βλέπετε λοιπόν πόσο πελώρες είναι οι επιπτώσεις. Ε, το δεύτερο σκέλος ε, της ερώτησης. Ε, πρέπει να ξέρουν και οι επιβάτες ποιες είναι οι διαδρομές και αν υπάρχει υπέρπτυση πάνω από πόλεμες ζώνες για να τους καθησυχάσουμε πιστεύουμε ότι η Ευρώπη ή ο κόσμος, ο Καό, έμαθε άλλες εδάγματα από τις ε, καταστροφές και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, τις γνώσεις μας για να επιτελέσουμε το καθήκον μας. Τον βοηθάει τον επιβάτη να ξέρει, να γνωρίζει τη διαδρομή. Ε, αμφιβάλλω, διότι ακόμη και στον αέρα αλλάζουν οι διαδρομές ε, και εμφανίζονται περιορισμοί και αλλάζει, αλλάζουν οι περιστάσεις. Ε, ε φανταστείτε, πτήση 10, 11, 12 ώρες. Είναι εν εξελίξη η διαδρομή, διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες και ο επιβάτης ε, ε ούτως ή άλλω βλέπει στην οθόνη που πάει το αεροπλάνο. 90% των αερομεταφορέων δείχνουν τη διαδρομή του. Ξέρει δηλαδή. Ε, γνωρίζει τη διαδρομή και νομίζω ότι πιο πολύ θα φέρει σε σύγχυση και θα, ε, θα, θα θορυβήσει τους επιβάτες ε, η κοινοποίηση της ε, διαδρομής. Πιστεύουμε ότι ε, η διαδικασία λειτουργεί χωρίς προβλήματα. Εάν υπάρξει αίτημα ε, να κοινοποιούνται αυτά τα δεδομένα, μπορούμε να το εξετάσουμε, αλλά φυσικά υπάρχει από την άλλη πλευρά η επιχειρηματολογία για τα μέτρα ασφάλειας. Μπορεί και κάποιοι άλλοι που δεν πρέπει να γνωρίζουν τη διαδρομή να τη γνωρίζουν και να τη χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Για το ζήτημα τη ε, στρατηγικής προσέγγιση για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό. Ιδιαίτερα για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό έχουμε συγκεκριμένους στόχους ε, και στα πλαίσια του περιβάλλοντος. Υπάρχουν συναντήσεις σε διεθνές επίπεδο επίσης ε, ε, και στα πλαίσια της ΙΚΑΟ θα γίνει μια συνέλευση σε δύο εβδομάδες για τη μείωση του, της χρήσης των υδρογονανθράκων Έχουμε συγκεκριμένους στόχους μέχρι το 2020, θα πρέπει οι στόχοι αυτοί να εκπληρωθούν και να γίνουν αναπόσπαστο τμήμα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και της νομοθεσίας που διέπει ε, τη λειτουργία του Eurocontrol. Η στρατηγική της Επιτρόπου Μπούλτς ε, λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον, Νομίζω όμως ότι περαιτέρω εκλεπτισμένες και περαιτέρω λεπτομέρειες σε επίπεδο νομοθετικό είναι απαραίτητες. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε κυρίως από το 2019 και μετά. Έχουμε εμείς καταρτήσει την λευκή βίβλο για το τι μένει να βελτιωθεί. Εγώ μπορώ να προσκαλέσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, είναι πολύ κοντά σας το Eurocontrol, να μας επισκεφθείτε με μεγάλη χαρά θα σας δείξουμε και ε, το κέντρο λειτουργίας μας, όπου συλλέγουμε όλα τα στοιχεία, τα επεξεργαζόμεθα και μπορούμε να σας δείξουμε το πώς τα χρησιμοποιούμε γενικά. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός ουρανός λοιπόν έχει ανάμεσα σε άλλους στόχους την ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνολογίας, οι ρυθμίσεις οι οποίες απαιτείται να γίνουν και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι εξοπλισμοί οι οποίοι απαιτούνται είναι πάρα πολύ φυσικά, έχουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος. Βέβαια η απόσβεση γίνεται με την έννοια ότι η χρήση τους μπορεί να ξεπεράσει και τα 20 χρόνια στη συνέχεια. Είμαστε υπερήφανοι για τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε, κανένας δεν έχει τέτοιου είδου μέσα Μιλάμε για τεχνολογίες ε, οι οποίες είναι ψηφιακού τύπου, ακόμα και το λεγόμενο Remote Tower Technology, το οποίο έχουμε το RTT, με ένα ιονή πύργο ελέγχου. Ξέχασα ένα σημείο, ίσως τα είπα πάρα πολύ γρήγορα, η συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά όργανα. Έχουμε μια συμφωνία υψηλού επίπεδου με την Ευρωπαϊκή Ένωση που περιγράφει λεπτομερώς την συνεργασία μας. Συνεργαζόμαστε επίσης με την ΕΑΣΑ Στα πλαίσια του, αλλά, της αλλαγής του κανονισμού της ΕΑΖΑ, θυμίζω ότι η ΕΑΣΑ είναι ο μηχανισμός επίβλεψης των συνθήκων ασφαλείας στον τομέα των αερομεταφορών και οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις συγκεκριμένες προσπάθειες που γίνονται στην ΕΑΣΑ. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υποστηριχθούν κάποιες ιδέες οι οποίες υπάρχουν για την απόκτηση από πλευρά της ΕΑΣΑ λειτουργικών ιδιωτήτων. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε εμείς να καλύψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και η Άσα είναι εκεί για να ελέγχει αν εκπληρούμε γενικά την αποστολή μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπρένερ για μια ακόμη φορά για τις εξηγήσεις σας και για την απάντηση που δώσατε σε όλες τις ερωτήσεις. Bueno, Περνάμε στο τελευταίο σημείο. Εμείς το 2011 είχαμε, προτείνει, είχαμε δώσει την έγκρισή μας για την διεύρυνση της συνεργασίας με το Ουσβεκιστάν στον τομέα της υφαντουργίας αλλά με ρήτρες ειδικέ για την παιδική εργασία και είχαμε κάνει και παραπομπές στην εμπορία και παραγωγή βάμβακος στο Πακιστάν. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Η ίντα θα ψηφίσει στις 9 και 10 Νοεμβρίου για τη διεύρυνση της συμφωνίας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λούνατσεκ, η οποία είναι η συγγήτρια. Ευχαριστώ και θα σας τα πω τώρα στα αγγλικά, λέει η κυρία Λούνατσεκ. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλώς ήρθατε στα Φρανία. Όπως θα ενθυμίστε, ήδη το 2011 το Ευρωκοινοβούλιο δεν συνήνεσε στην παράταση ισχύω της συμφωνίας λόγω αναφορών που υπήρχαν για παιδική εργασία και αναγκαστική παιδική εργασία και τα είχαμε περιλάβει αυτά και στην θέση μας του Απριλίου 2016 ως Κοινοβούλιο ότι δεν θα εγκρίνουμε εάν δεν αντιμετωπιστεί και εξαλειφθεί η παιδική εργασία και στο εθνικό και στο τοπικό επίπεδο. Είδαμε διαμέσου των ετών ότι λόγω τη έλλειψη εγκρίσεω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βεβαίω και λόγω τη αντιδράσεως και άλλων θεσμικών οργάνων και τη Παγκόσμια Τράπεζα και του, Παγκόσμιου, ε, του μάλλον Οργανισμού εργασία κλπ. Πιέστηκε το Ζουμπικιστάν να προχωρήσει στο θέμα αυτό και να αρχίσει να μειώνει την παιδική εργασία και βέβαια την καταναγκαστική εργασία. Για την παιδική εργασία είδαμε πράγματι σημαντικά βήματα πρόοδου. Είναι γεγονό τώρα ότι η παιδική εργασία αντιμετωπίζεται και εκεί ως κοινωνικά ανεύθυνη υπόθεση. Βεβαίως μπορεί να συμβαίνει ακόμα. Ε, διεξήχθηκε ακρόαση στην ε, αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, για την καταναγκαστική εργασία υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις, όμως κατά την άποψή μου, αλλά και τα ίδια λένε και πολλοί από τον ILO, αλλά και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες που δεν του επιτρέπεται στην πραγματικότητα καν να παρακολουθούν τις υποθέσεις αυτές στην ίδια τη χώρα. Μου είπαν πάντως ότι υπάρχουν ε, αναφορές και στον τύπο και ότι για την εσοδεία που θα αρχίσει τώρα, ε, μεθαύριο, Υπάρχουν ειδήσει λοιπόν που ε, λένε ότι αναγκάζουν και δημοσίους υπαλλήλου και γιατρούς και άλλους να πάνε να δουλέψουν στην ε, συγκομιδή και αν δεν το πράξουν αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να τους επιβληθούν πρόστιμα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο προτείνω στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να μην εγκρίνει πριν να λάβουμε είδηση ότι η συγκομιδή που θα αρχίσει τώρα στις 10 Σεπτεμβρίου, ο Άιελό μας είπε πριν ότι θα δώσει τελική μορφή πλέον στις εκθέσεις του ε, Δεκέμβριο ή αρχές Ιανουαρίου, άρα ίσως έχουμε κάποιες πρώτες τοποθετήσεις τον Δεκέμβριο και εδώ έρχεται το δεύτερο θέμα τώρα. Απεβίωσε προ λίγων ημερών ο πρόεδρος Καρίμοφ. Δεν είναι σαφής η πολιτική σκηνή και πώς θα εξελιχθεί το πολιτικό τοπίο στο Ουσμπεκιστάν. Ως κοινοβούλιο μπορούμε να ασκήσουμε μεγαλύτερη πίεση διότι πίεση σημαίνει και μεγαλύτερη πίεση για εκδημοκρατισμό της χώρας. Θυμάστε τη σφαγή το 2005 με πολλές εκατοντάδες νεκρών και τραυματιών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε είχε επιβάλει διπλού είδους κυρώσεις σε βάρος της κυβέρνησης του Ουσμπεκιστάν και προξενικές θεωρήσεις και οικονομικές κλπ. Οι μη κρατικέ οργανώσεις τότε είχαν ωστόσο ασκήσει κριτική, αργότερα δηλαδή, όταν ανέστρεψε την θέση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γνωρίζουμε τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος Ακούμε ότι ίσως αναλάβει ο νυν πρωθυπουργός. Είναι είναι, είναι σωστό νομίζω να μην δοθεί τώρα η συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ζητήσουμε η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να βελτιωθεί σημαντικά πριν να δώσουμε την ε, συνένεση, διότι αυτό εντάσσεται και στην PCA, στο άρθρο 2 της οποίας λέγεται καθαρά ότι η PCA απαιτεί από τα συμβαλόμενα μέρη να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και προφανώς δεν σημαίνει αυτό. Ο Βυσιόγεφ που είναι ο νυν Πρωθυπουργό και που ίσως να διαδεχθεί στην Προεδρία των Καρίμοφ είναι και αρμόδιος για τη Γεωργία. Και είναι αυτός ο οποίος έχει επιβάλει ποσοστώσεις και στις τοπικές κυβερνήσεις για τη συγκομιδή του βαμβακιού. Έχω συζητήσει και με, τις κοιόδης, με τους και λόγω του, της μετάβασης, πολιτικής μετάβασης αυτή τη στιγμή στο Ουσβεκιστάν και λόγω ε, των άλλων εξελίξεων να μην, να μην δώσουμε τώρα την έγκρισή μας. Δεν είμαι απολύτως αντίθετη να δοθεί έγκριση. Νομίζω όμως ότι είναι ένα μέσον πιέσος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα για να επιτύχουμε αυτά που, να υλοποιηθούν δηλαδή αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί. Και έχει δεσμευτεί και η κυβέρνηση του Ουσβεκιστάν. Προτείνω λοιπόν συνάντηση των σκιωδών εισηγητών την επόμενη εβδομάδα, ώστε να μπορέσουμε να μορφώσουμε άποψη γι' αυτό και να συντάξουμε την ομοδότηση. Ευχαριστώ από τότε που ο Κουκάν, που είναι εισηγητή και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, δεν μπορούσε να έρθει σήμερα, μου ζήτησε να διαβάσω την δήλωσή του. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας είναι κάτι το κρίσιμο. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει ξεχωριστά σε κάθε χώρα βέβαια. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με το Ουσμπεκιστάν. Είδαμε την έκθεση του φθινοπόρου του 2015 ε, της υπηρεσίας της, ε, του ILO Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα παιδικής εργασίας και μπορεί να συμπεριληφθεί η, η φαντουργία στη συμφωνία. Α, το, ε, η χώρα αυτή δεν, έχει, δεν είναι μέλος ε, του ΠΟΕ και γι' αυτό θα ήθελα να συμφωνήσω με τη διαδικασία σύμφωνης γνώμης που προτείνει η ΙΝΤΕ. Πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να το συζητήσουμε αυτό ελπίζοντας να ψηφίσουμε τελικά το Δεκέμβριο. Άκουσα και τα διάφορα επιχειρήματα της κυρίας Λούνατσεκ. Θα ήθελα να πω ότι ο κύριος Κουκάν πιστεύει ότι η ΑΦΕΤ δεν είναι η αρμόδια επιτροπή, ε, επί της ουσίας εννοώ, και θα συμφωνήσω και εγώ μαζί του ότι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή πρέπει να αναλάβει την πρωτοβουλία έγκρισης. Ευχαριστώ. Πράγματι είμαι εισηγήτρια για το θέμα αυτό στην Επιτροπή Ίντα. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε, λέει η κυρία Ρενά, στο θέμα. Η κυρία Λούνατσεκ έκανε, μας έδωσε ένα μικρό ιστορικό των σχέσεών μας με το Ουσβεκιστάν. Είναι ένα θέμα που γνωρίζουμε εδώ και αρκετό καιρό. Υπάρχει ήδη μια συμφωνία εταιρική από το 1999 με την συγκεκριμένη χώρα Νομίζω ότι τα επιχειρήματα τα οποία εξέθεσε η κυρία Λούνατσεκ θα μπορούσαν να θέσουν σε αμφισβήτηση το σύνολο της σχέσης συνεργασίας με την συγκεκριμένη χώρα. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για μας να ξεκινήσουμε μια τέτοια δυναμική συνεργασίας. Είναι μία από τις λίγες χώρες της περιοχής που μπόρεσε να ανοίξει κάπως ε, τις διαδικασίες του. Κάνουμε πάντα κριτική στις, δημοκρατικές, στις προσπάθειες για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, αλλά προσπάθησε να συνεργαστεί μετά από πιέσεις του Κοινοβουλίου ε, και συνεργάστηκε με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας επίσης. Το να στείλουμε ένα αρνητικό μήνυμα στο Ουσμπεκιστάν, ενώ έχει επαναλαμβάνω συνεργαστεί, έχει ανοιχτεί ε, νομίζω ότι θα ήταν ένα κακό, μα κακό μήνυμα. Αντίθετα αυτό το οποίο ζήτησα από την ίντα είναι να προσπαθήσουμε να συνδέσουμε με την απόφαση επικύρωσης του πρωτοκόλου για το Βάμβακα και ένα ψήφισμα το οποίο θα μας επιτρέψει να δώσουμε αν θέλετε και τη δική μας εικόνα για την κατάσταση στο Ουσμπεκιστάν και θα μας επιτρέψει να ενημερώσουμε σωστά το Ουσμπεκιστάν ε, για το τι περιμένουμε ακόμα περισσότερο να γίνει στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν εγώ ε, συμφωνώ με τα επιχείρηματα της κυρίας Λούνατσεκ. Προφανώς η κατάσταση δεν είναι ιδανική. Όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο Ουσμπεκιστάν το μαρτυρούν αυτό όταν έχουν την δυνατότητα να το κάνουν Απ' την άλλη όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και δεν πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα κλεισίματος της Ευρώπης προς τη χώρα αυτή, ενώ η κατάσταση βελτιώνεται. Έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά σε επίπεδο της ΣΥΝΤΑ με τους διάφορους συνομιλητές μας. Συναντηθήκαμε και με τα ουσμπεκικά συνδικάτα και στον τομέα της παιδικής εργασίας και στον τομέα της καταναγκαστικής εργασίας Νομίζω ότι μιλήσαμε και με την κυβέρνηση βέβαια, είχαμε και μια κοινή ομάδα εργασίας με το Διεθνές Γραφείο, το οποίο μας έχει περιγράψει θετικά τις αλλαγές τα τελευταία χρόνια, τρία χρόνια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και μια νέα αποστολή του ΟΗΤΕ, του Διεθνούς Γραφείου, κατά τη διάρκεια της συλλογής της νέας εσοδείας Βάμβακα, και νομίζω ότι οι ε, αναφορές ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Ίσως να υπάρξουν πολιτικές αλλαγές στο Ουσμπεκιστάν τις επόμενες εβδομάδες. Αλλά αντί να κλείσουμε τις θέσεις μας, να κλειστούμε μάλλον, νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε ευρωπαϊκά ανοίγματα στις πολιτικές αλλαγές οι οποίες μπορεί να επισυμβούν στην χώρα αυτή. <clears throat> θα λάβουμε υπόψη μας αυτά τα οποία θα πει η γνωμοδότηση ΑΦΕΤ για την επικύρωση του προκόλου για το βαμβάκι. Η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε και σε σχέση με τις βελτιώσεις οι οποίες έχουν γίνει αλλά και με τις απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Έχουμε ένα παράδειγμα εδώ για το τι σημασία έχει η στρατηγική και πολιτική θέση μιας χώρας. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε γενικά να συνεχιστεί η διαδικασία και φυσικά έχει μεγάλη σημασία και η γνώμη των ανθρώπων οι οποίοι έχουν αμφιβολίες αλλά νομίζω ότι στα πλαίσια της συνεργασίας ε, θα ήθελα να πω στην κυρία Λούνατσεκ που πιστεύει ότι δεν πρέπει να διευρυνθεί η συμφωνία αυτής της συνεργασίας Νομίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα ήθελα ε, δεν θα ήθελα να χρησιμοποιούν βαμβάκι το οποίο να προέρχεται από τα χέρια δούλων. Ε, Ευχαριστώ. Η δική μου πρόταση θα έχει ως εξής. Η είναι η αρμόδια της Εγώ πήρα το λόγο ο ίδιος πριν να, τον, ε, πριν να μιλήσει η Λούνατσο. Περιμένετε λοιπόν μέχρι να τελειώσω. Η ΙΝΤΑ λοιπόν είναι η αρμόδια επιστοσίας επιτροπή. Την ακούσαμε την άποψή της. Που στοχεύει στο να περιληφθούν και τα υφαντουργικά μέσα στη συμφωνία. και η ίντα είναι διατεθειμένη να δεχθεί ψήφισμα στο οποίο να περιλαμβάνει και τις κριτικές μας τοποθετήσεις απέναντι στην κατάσταση των δικαιωμάτων στο Ουσβεκιστάν. Η πρότασή μου λοιπόν είναι να ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα της ίντα με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν σύντομα προτάσει ήδη την εβδομάδα αυτή για τη γνωμοδότηση και μέχρι τις 26 ενάτου, 18 ε, βραδινές ώρες, να έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε τροπολογίες. Και να δούμε μετά πώς θα προχωρήσει. Δέχεστε τη διαδικασία αυτή η κυρία Συγγήτρια της Επιτροπής Εξωτερικών. Λούνατσεκ. Ευχαριστώ για την πρότασή σας. Έχοντας ακούσει τους συναδέλφους και βεβαίως και την εισηγήτρια της ΣΥΝΤΑ και τους σοσιαλδημοκράτες, έχω ωστόσο να κάνω, μάλλον να επαναλάβω την πρόταση που έκανα πριν και για την κυρία Αρενά. Δεν θέλω να μπλοκάρω την έγκριση από το Κοινοβούλιο. Θέλω να δοθεί η έγκριση. Η επιθυμία μου, το αίτημά μου είναι να περιμένουμε ένα μήνα ώστε να μπορέσει ο ILO να υποβάλει την έκθεσή του τον Δεκέμβρη. Γνωρίζω ποια είναι η απόφαση της ΣΥΝΤΑ. Αντιλαμβάνομαι ότι, και το εκτιμώ ότι η ΙΝΤΑ δέχθηκε να συνταχθεί ψήφισμα Άκουσα τι είπε ο Πρόεδρος και υποθέτω ότι προς τα εκεί θα κινηθούμε εν τέλει. Παρ' όλα αυτά επιμένω να γίνει συνάντηση και οδόν εισηγητών την επόμενη εβδομάδα και εν τέλει ε, θα βρεθώ και εγώ σύμφωνη, αλλά για πολιτικούς λόγους νομίζω ότι η συνένεση είναι μεν σημαντική, η έγκρισή μας δηλαδή είναι σημαντική, αλλά πρέπει να περιληφθούν οι διατυπώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα για ζητήματα δημοκρατίας και ιδίως τώρα μετά τον θάνατο του Προέδρου και όπου κανείς δεν γνωρίζει πώς θα διαμορφωθεί η πολιτική σκηνή στο Ουσβικιστάν στο προσεχές μέλλον. 26 Ιανουαρίου λοιπόν. Έχουμε χρόνο αρκετό για να γίνουν προτάσεις. θα ακολουθήσουμε το χρονοδιάγραμμα της ίντα, θα συνεχίσουμε να συζητούμε μαζί τους. Θα έχουμε και τη δυνατότητα να συνεργαστούμε την επόμενη εβδομάδα και προτείνω να θυρίσετε το χρονοδιάγραμμα που σας ανέπτυξα προηγουμένως. και να παραμείνουμε σε διασύνδεση με τις ε, εργασίες της ΣΥΝΤΑ ώστε να ολοκληρώσουμε έγκαιρα. Όμως, τώρα, πριν να κλείσω, με μεγάλη μας χαρά βλέπω μεταξύ μας την Άντια Σαρτσένκο. Ε, just ε, Μόλις συναντήθηκα δίμερος μαζί της και εξέφρασα τη γνώμη ότι Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που την βλέπουμε εδώ κοντά μας, εν ειρήνη και σε καλή υγεία. Και τη είπα ποτέ πια απεργία πείνας. Θα θέλαμε να σας έχουμε όπως είστε. Θέλει να ευχαριστήσει για το γεγονός ότι πολλοί ευρωβουλευτές αγωνίστηκαν για την ελευθερία της και αν θέλετε να σας δώσουμε λίγα λεπτά το λόγο Είμαι, είμαι πολύ ευγνώμων για τις ε, προσπάθειές σας. Είδατε ότι μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική ζωή ενός προσώπου. Είμαι βεβαία και πιστεύω και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο τόπος εκείνος όπου γίνονται σεβαστές οι αξίες της ανθρώπινης ζωής και της αξιοπρέπειας του καθενός. Ευχαριστώ πολύ. Ich danke Ihnen Ασφαλώς θα έχετε την υποστήριξή μας και στο μέλλον, στην περίπτωση της Ουκρανίας, θα αγωνιστούμε για το απαραβία, υπέρ του απαραβίαστου της επικρατείας της Ουκρανίας για την πάυση των εχθροπραξιών και θα πράξουμε ό,τι μπορούμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως πράξαμε ως τώρα, για να βοηθήσουμε με την ελπίδα άλλωστε η Ουκρανία να βρει την δύναμη να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία, την δημοκρατία, να ενισχύσει τον αγώνα κατά της διαφθοράς και με τον τρόπο αυτό να εμφανιστεί πιο ισχυρή απέναντι σε αυτή την ρωσική επιθετικότητα που ζήσαμε. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας εύχομαι κάθε τι το καλό και προσωπικά. Λίγη συνεδρίαση.